Welcome Καλώς ορίσατε. Να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας σήμερα. Έχουμε βεβαρημένη ημερήσια διάταξη. Votes ε, for, for Έχουμε τέσσερις εκθέσεις να ψηφίσουμε και πρέπει να ξεκινήσουμε αν και έχουν καθυστερήσει κάποιοι συνάδελφοι, διότι λόγω κάποιου εκτακτού συναγερμού έχουν ε, ε, κλείσει οι δρόμοι. Ε, Ξεκινάμε με το σχέδιο γνωμοδότηση της Αμπέν Χεράη για την φορητότητα των, του διαδικτυακού περιεχομένου. Αν έχετε τις κάρτες σας μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσω. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 98, υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 99, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 117. Μακλάρκινγκ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για πάμε πάλι υπέρ για την 121, κατά, αποχές, απορρίπτεται μάλλον, 120 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 122 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 123 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 124 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 125 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 126 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 127 υπέρ, κατά, Υπέρ και πάλι εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 στο άρθρο 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 στην επόμενη σελίδα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 στην επόμενη σελίδα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία... Α, συγγνώμη. 17 της εισηγήτριας, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Που είναι ταυτόσιμη με την 156. Συμβαστική τροπολογία 10, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 22, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 36 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13 στην επόμενη σελίδα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 15, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 16, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 71, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 72, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 73, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 74 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 75 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 18, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 84, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία στο σχέδιο γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. 25 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια στη συντάκτρια της γνωμοδότησης. Πολύ σημαντική και ευχαριστώ και τους κοιόδης συντάκτες για τη δουλειά τους. Θα συνεχίσουμε τώρα με το σχέδιο γνωμοδοτήσεως του Στέφανο Μαούλου. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ως εξής. Τροπολογία 8 στο πρώτο άρθρο. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41. Όχι, με συγχωρείτε, 40, 40 λέει η 40 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή τροπολογία 10 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμών 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 στο κάτω μέρος της σελίδος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ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 κατά αποχές απορρίπτεται και αυτό 25 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 εισηγήτου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά απο... δεν λέει αποχές πρόεδρος εγκρίνεται με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Απορρίπτεται, λέει η πρόεδρος. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. 16 ψήφοι υπέρ, 14 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 εισήγητου υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία επί του σχεδίου, αρχίζει η ψηφοφορία, είναι ε, ονομαστική, πέρας. ψήφι 20 υπέρ, 7 κατά και 3 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση. Συγχαρητήρια κύριε Μαούλου. Και ευχαριστώ βεβαίως και, στους, και τους συζητητές. Και ακολουθεί η επόμενη για τον προϋπολογισμό του 2017 και εντολή για τριμερή διάλογο είναι η, το σχέδιο μάλλον του κυρίου Σδρογεύσκη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 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 με συγχωρείτε, εδώ ζητείτε κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30. Η τροπολογία 30. Πάλι ζητείτε εδώ ξεχωριστή, μάλλον δηλαδή ξεχωρία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Εδώ θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, όπως είπα. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν 18 υπέρ 12 κατά. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 28 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ομοίως. Παρέμβαση χωρίς ε, μικρόφωνο. 31. Την ψηφίσαμε. Τώρα είμαστε στην 33. 33 λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Με συγχωρείτε, όχι, εδώ ζητείτε, έχει ζητηθεί ψηφοφορία κατά τμήματα από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Πρώτο τμήμα λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 του συγγετού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές εδώ θα κάνουμε επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία επί του συνόλου της ε, γνωμοδοτήσεως. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Ωραία, τώρα λίγη ψηφοφορία. 24 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Σδρογεύσκη. Αλλά ο κύριος Δρογεύσκη δεν, ε, τελειώσαμε. Υπάρχει και μια άλλη γνωμοδότηση, στρατηγική ανακοίνωση της Ένωσης ως απάντηση στην προπαγάνδα από τρίτους εις βάρους της. Ας αρχίσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11, υπέρ, κατά, αποχές. Ας ελέγξουμε καλύτερα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Ακατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ.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 Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 35, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 κατά τμήματα όπως η η άλλη. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά αν θέλετε. 38 πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Πέρας. 21 ψηφοί υπέρ, 9 κατά. Θέλετε να ελέγξουμε και το δεύτερο. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40. Κατά τμήματα, όπως ζήτησε το ΕΛΚ το και η ΑΛΤΕ. Υπέρ. Πρώτο τμήμα μάλλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49. Κατά τμήματα, όπως ζήτησε το ΕΛΚ, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 16 υπέρ, 14 κατά εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. A υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας με 25 ψήφους υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια στον κύριο Στρογεύσκη. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία για σήμερα. Και... Και θα πρέπει τώρα να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε με το επόμενο θέμα.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 Bene. Welcome to... Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Έχουμε εδώ την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Κλέρ Μπιούρι, αναπλώτρια γενικά διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Connect και τη τμήματάρχη του τμήματος Connect, της Γενικής Διεύθυνσης Connect. Σας ευχαριστούμε πολύ και χαιρόμαστε για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί του ζητήματος μαζί σας. Θα συνεχίσω στα Ιταλικά, αν μου επιτρέπετε. Τα λέω καλύτερα στα Ιταλικά. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν ότι σήμερα θα κάνουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της Επιτροπής μας. Είμαστε και ε, αρμόδιοι, έχουμε την πλήρη αρμοδιότητα και θα ήθελα να πω ότι σαφώς ε, και ε, βρισκόμαστε και σε ένα πάρα πολύ σημαντικό στάδιο για τα όσα έχουμε σήμερα στο σύστημα των οπτικοακουστικών μέσων, όχι μόνο των τηλεοράσεων, αλλά και τη μεγάλη σύγκληση που υπάρχει μεταξύ τηλεοπτικής μετάδασης και ε, μεταδόσεων μέσω διαδικτύου. Ε, έχουμε περιεχόμενο πλέον on demand, ε, πρόσβαση από ε, κινητές ε, και σταθερές συσκευές και παρά το γεγονός ότι η παραδοσιακή ραδιοτηλεόραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόμα ισχυρή παρουσία, το καταδεικνύουν αυτό και τα στοιχεία, Υπάρχουν όμως και νέα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία αναδύονται διαδικτυακά, αν και ε, δεν είναι πάντα στην επιθυμητή ε, κατάσταση που θα θέλαμε εμείς, δηλαδή με ισότιμους όρους ανταγωνισμούς. Υπάρχει λοιπόν ε, αύξηση της διαδικτυακής δραστηριότητας, αυξάνονται οι μεταδόσεις, υπάρχουν πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, προσφέρουν οπτικό-ακουστικό περιεχόμενο διαδικτυακά και στοχεύουν φυσικά στο ίδιο κοινό. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο πρώτος ε, λόγος ε, για τον οποίο γίνεται αναθεώρηση αυτής της οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες είναι αυτή η ταχύτητα, ταχύτατη ε, αλλαγή η οποία κατά την άποψή μας πρέπει να έχει και πιο ομογενείς κανόνες ομοιογενείς κανόνες προστασίας όλων των φορέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της στις 25 Μαΐου ως τμήμα της ε, ψηφιακής στρατηγικής για την νέα αγορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ε, θα προτιμούσαμε να την αποκαλούμε Ευρωπαϊκή ε, Ψηφιακή Στρατηγική, διότι δεν αφορά μόνο την αγορά, αλλά και τους πολίτες και τους χρήστες, αλλά και το περιεχόμενο. Και πρόκειται φυσικά για μια πρόταση η οποία στόχο έχει να προσαρμόσει τους κανόνες σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε κάποια θέματα, παραδείγματο χάρη την επέκταση και στα διαδικτυακά ζητήματα των υποχρεώσεων, αλλά και θέματα προστασίας ε, για τους ανηλίκους, ε, για τη ρητορία μίσους ε, και ακόμα και την πρόκληση σε βία ή σε μίσος. Να υπάρχει κατάλληλη προστασία για αυτές τις πλατφόρμες Υπάρχει και ένα σχετικό ad hoc κεφάλαιο που αφορά τα θέματα αυτά, αλλά θα πρέπει να δούμε και ποιες πλατφόρμες ε, αφορούν αυτή την οδηγία και τι εξαιρείται και θεωρείται τμήμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ε, διότι θεωρούμε ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο σε αυτές τις πλατφόρμες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να υπάρχει κατάλληλη προστασία ε, και κατάλληλα κίνητρα για παραγωγή και διανομή ενός ε, ποσοστού ευρωπαϊκών έργων. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανεξάρτητες παραγωγές. Υπάρχει φυσικά το θέμα της ε, εμπορικής ε, επικοινωνίας. Υπάρχει νομοθεσία και σχετικά άρθρα που καλύπτουν τη διανομή με διαφορετικό τρόπο και την ευελιξία, αν θέλετε, για τα εμπορικά ζητήματα. θέματα στα οποία θα εμβαθύνουν φυσικά και οι αρμόδιοι συγητέ και οι ισχυώδει συγητέ και υπάρχει και το θέμα της πρόσβασης φυσικά, το οποίο θα σχολιάσουν αργότερα συνάδελφοι. Πριν ε, ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση όμως, θα ήθελα να υπενθυμίσω, διότι την περασμένη εβδομάδα ε, είχαμε και κάποια ευαίσθητα τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν και στον τύπο, στην πραγματικότητα σε μία εφημερίδα μόνον, και αφορούν ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για μας ε, και ε, πρέπει να γίνει και κατάλληλη επαλήθευση και να το συζητήσουμε ανοιχτά. Ε, θέματα δηλαδή που αφορούν την σύγκρουση συμφερόντων και θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους αρμοδίους εισηγητές. Να σας πω ότι εχθές το απόγευμα εμβαθύναμε όσο έπρεπε, κατόπιν αιτήματος φυσικά και διαφόρων πολιτικών ομάδων, αλλά θεωρούσα και εγώ την υποχρέωσή μας. Εμβαθύναμε λοιπόν στο θέμα αυτό στη συνεδρία των συντονιστών. Υπήρξε μια αναλυτική δήλωση ε, την οποία παρουσίασε η, συνάδελφη Πέτρα Καμερ, η συνάδελφος Πέτρα Καμερέβερτ ε, και επίσης και η συνάδελφος Φεράιαν ε, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και θεωρώ ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων και των πολιτικών ομάδων που εκπροσωπούσαν θεωρούν ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε, μπορούμε να συζητήσουμε τις διάφορες πολιτικές θέσεις, οι οποίες είναι καθόλου θεμητό να συζητούνται, αλλά η νομική βάση θεωρείται ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί δεν είναι ε, εύκολη η υλοποίηση και θεωρώ ότι καταλήξαμε όλοι στη σύμφωνη γνώμη ότι αυτό το προφίλ δεν ε, καλύπτει και αυτές τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Θα ήθελα να το επενθυμίσω εδώ, διότι ε, θεωρώ ότι εμείς θα πρέπει να ε, εγγυηθούμε και την τιμή των συναδέλφων που θα ασχοληθούν με τα θέματα αυτά που είναι τόσο σημαντικά και ότι ο καλύτερος τρόπος για να απαντήσουμε σε όλες τις μορφές ε, πιέσεων, ε, είτε πρέπει είτε δεν πρέπει να γίνουν. Αυτά υπάρχουν σε όλα τα κοινοβούλια, υπάρχει και στο δικό μα, αλλά θα πρέπει να εγγυηθούμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και εγώ χαίρομαι για τη μέθοδο που επέλεξαν να ακολουθήσουν οι συνεισηγητέ και οι σκιώδη εισηγητές να υπάρχει μία κοινή διαδικασία μαζί με όλους τους κοιόδης συζητητές ε, στις συναντήσεις με τους διαφόρους ενδιαφερομένους. Νομίζω ότι έχετε προβλέψει τρεις συνεδριάσεις οι οποίες θα είναι αφιερωμένες στις διάφορες κατηγορίες ενδιαφερομένων και εκεί θα συμμετέχουν όλοι οι σκιώδεις συζητητές Στις 26 του μηνός θα γίνει ακρόαση στην Επιτροπή Πολιτισμού με εμπειρογνώμονες για το θέμα αυτό και όλη η διαδικασία θα γίνει με πλήρη διαφάνεια και με συμμετοχή όλων των συναδέλφων. Αυτό γιατί πρέπει να προστατεύσουμε και το Κοινοβούλιο από οποιαδήποτε χειραγωγή και πρέπει να απαντήσουμε φυσικά ε, και να εγγυηθούμε ότι θα γίνουν όλα με απόλυτη διαφάνεια. Να υπάρχει διαφάνεια λόγω αυτών των εξωτερικών παρεμβάσεων και πιέσεων. Νομίζω ότι εδώ τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στις συναδέλφους ε, ε, που είναι οι συνεισηγήτριες, στη συνάδελφο Φεράιαν και συνέχεια στην κυρία Καμερέβερτ, οι οποίες σε πέντε λεπτά θα κάνουν κάποιες εισαγωγικέ παρατηρήσεις και από εκεί και πέρα θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στου συναδέλφους, στου κοιόδη και σε όποιον θέλει συναλλάβει το λόγο στη συνέχεια. Παρακαλώ, προτιμάτε να ακούσετε πρώτα την Επιτροπή, διότι η διαδικασία προβλέπει να μιλήσετε εσεί πρώτα. Δεν πειράζει, θα περάσουμε απευθεία στην παρουσίαση τη επιτροπή θα λόγο, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, που με καλέσατε σήμερα. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ μαζί σας, στην Επιτροπή σας, για να συνεχίσω τη συζήτηση η οποία άρχισε πριν από ορισμένους μήνες όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμαζε ε, τη, στα πλαίσια του κανονισμού ΡΙΦΗ την αναθεώρηση της οδηγίας για τα ακουστικά μέσα. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε μερικά εισαγωγικά σχόλια. Η ψηφιακή ε, ενιαία αγορά χρειάζεται μια στρατηγική. Η στρατηγική όμως αυτή δεν πρέπει να αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και τον τρόπο που επηρεάζει τις ζωές των πολιτών και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες θα χρησιμοποιούν τα μέσα ενημέρωσης, κάτι το οποίο αλλάζει με ταχύτητα τους ρυθμούς αυτή την εποχή είναι μία μετάβαση που θα γίνει σταδιακά. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μία επιτάχυνση. Από την παραδοσιακή ραδιοτηλεόραση στον, στην ε, επιγραμμική Νομίζω πως ε, δεν πρόκειται εδώ για κάποια επανάσταση, αλλά για εξέλιξη. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε το εφιστάμενο πλαίσιο έτσι ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα ε, και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών οι οποίοι χρησιμοποιούν ε, περιεχόμενο οπτικοακουστικών μέσων. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως πρέπει να κοιτάξουμε με προσοχή τον, ε, την ε, οδηγία και να κρατήσουμε τα στοιχεία που είναι χρήσιμα, να αναθεωρήσουμε όμως και να αλλάξουμε τα στοιχεία που πρέπει και είναι παροχημένα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, λάβει κάποια, ε, έχει κάνει κάποια γενναία βήματα, υπάρχουν κάποιες διατάξεις τις οποίες θεωρούμε παροχημένες και χρειάζονται αλλαγή. Γίνονται όμως κάποιες σημαντικές αλλαγές, τουλάχιστον αυτό προτείνουμε οι οποίε αλλαγέ θα μας βοηθήσουν να λάβουμε υπόψη τα νέα δεδομένα και τους νέους ε, ε, φορεί και παρόχους ε, περιεχομένου για τους πολίτες μας. Τώρα θα ήθελα αρχικά να σας τονίσω τα ουσιώδη στοιχεία και τις βασικές καινοτομίε πρώτο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι πώς διατηρείται η ε, αρχή της χώρας προέλευσης. Αυτό είναι κάτι που έχει αντέξει στον χρόνο και θα βοηθήσει ε, τους ε, φορείς ερωτηλεόρασης να εκπέμπουν περιεχόμενο σε άλλα κράτη-μέλη. Αν δούμε τα νούμερα θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα περιεχομένου από μία χώρα, από ένα κατός μέλος στο άλλο και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όσους ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό και για το περιεχόμενο και είναι και καλό για τους πολίτες επίσης. Ωστόσο, θα θέλαμε η αρχή λειτουργίας να γίνει πιο απλή. Είδαμε ότι στην πορεία πολλές φορές συναντήσαμε δυσκολίες για το πού ε, εδεύει ένας ε, πάροχος, σε ποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε λοιπόν οι ρυθμιστικές αρχές να έχουν λίγο ευκολότερη ε, δουλειά στον εντοπισμό της έδρας ενδεχομένως να υπάρχουν ορισμένες εθνικές ιδιαιτερότητες, ενδεχομένως να υπάρχουν περιορισμοί, όμως πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν, αντί να αμφισβητήσουμε την αρχή της ε, χώρας προέλευσης, κάτι το οποίο ακούσαμε κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, ε, θεωρούμε με συντριπτική πλειοψηφία ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, πως έχει λειτουργήσει πολύ σωστά μέχρι τώρα. Γι' αυτό λοιπόν προτείναμε απλούστευση, επεξήγηση, με, τον, ε, με τρόπο έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να υποφεληθούν περισσότερο από αυτό. Τώρα, ω προ τι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σχετικά με την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, ε, είναι κάτι το οποίο θα ε, επαναξεταστεί. Αυτά λοιπόν για την αρχή τη χώρα προέλεύση. Τώρα, καινοτομίε. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω πω αναφερθήκατε στην ανάγκη να υπάρχει μια ισορροπημένη πρόταση και πώ λοιπόν θα προσαρμοστούμε στι ε, αλλαγέ τη αγορά. Καταρχάς, προτείνουμε να δοθεί περισσότερη ευελιξία στους ε, ε, στους ε, φορείς ραδιοτηλεόρασης σχετικά με τις διαφημίσεις. Έχουν αλλάξει πλέον οι καιροί και πολλοί χρήστες πιο γρήγορα και πιο εύκολα αλλάζουν μέσο Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλέ φορέ στο διαδίκτυο υπάρχει περιεχόμενο χωρί διαφημίσει και πώ οι χρήστε προτιμούν ε, να βλέπουν κάτι από την αρχή στο τέλο παρά να υπάρχουν διακοπέ για διαφημίσει. Υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό αυτή τη στιγμή ε, ω προ το εισόδημα από διαφημίσει. και με το εισόδημα αυτό μπορούν φυσικά να ε, δημιουργούν περιεχόμενο το οποίο θα κάνουν διαθέσιμο για τους χρήστες. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να τροποποιηθεί το όριο των 12 λεπτών ανά ώρα, του 20% δηλαδή, και να δοθεί περισσότερη ευελιξία, η οποία θα εφαρμόζει την αρχή του 20% από τις 7 το πρωί στις 11 το βράδυ. Με αυτόν τον τρόπο, οι ρεδοτηλεοπτικοί φορείς θα μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι πού θέλουν να ε, ρίξουν τις περισσότερες διαφημίσεις και πού θέλουν να ε, προσελκύσουν το περισσότερο εισόδημα από διαφημίσεις. Θα υπάρχει δηλαδή ενδεχομένως ε, μεγαλύτερο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιήσουν για δημιουργία περιεχομένου. Έπειτα, ε, ενίσχυση κανόνων για τις υπηρεσίες on demand, κατόπιν ζήτηση. Νομίζω πως και εσείς κυρία Πρόεδρε μας είπατε ότι αυτές οι υπηρεσίες on demand έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Χρειάζεται φυσικά να προσέξουμε τους κανόνες για την προστασία ανηλίκων, έτσι ώστε αυτοί να ευθυγραμμίζονται με ε, τους ρεδιοτηλεοπτικούς φορείς. Φυσικά, έχουμε προτείνει ένα ελάχιστο ποσοστό ε, περιεχομένου on demand και προτείνουμε τα κράτη-μέλη να μπορούν να ε, επιβάλλουν οικονομικές ε, εισφορές από τις υπηρεσίες on demand και εκείνες οι οποίες ε, προέρχονται από κάποιο άλλο κράτος μέλος. Όπως σας είπα, δεν πρόκειται για επανάσταση αλλά εξέλιξη. Σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν κανόνες που ορίζουν ένα ποσοστό πάνω από το 20%, όμως αυτό που θέλουμε εμείς είναι μία συνεχόμενη και συνεπής συνεισφορά προς το περιεχόμενο. Τέλος, ε, τελευταίο καινοτόμο στοιχείο, ίσως και από τα πιο σημαντικά, ίσως και το σημαντικότερο, έχει να κάνει με τις πλατφόρμες ανταλλαγής περιεχομένου, το video sharing, οι οποίες αυτή τη στιγμή ε, καλύπτονται από την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα, για τους ίδιους λόγους με τις προηγούμενες. Μας αναφέρετε, κυρία Πρόεδρε, την διασύνδεση με την οδηγία για το ηλεκτρονικό περιεχόμενο και αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να συμπληρώσουμε την οδηγία αυτή, να μην δηλαδή να τρέψουμε τους κανόνες της, διότι θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ σημαντική για την καινοτομία, αλλά να καταστεί σαφές ότι πρέπει να υπάρχει κάποια υποχρέωση για αυτές τις ε, πλατφόρμες να υπάρχουν κάποια, ε, κάποια μέσα, κάποιες ρυθμίσεις που θα προστατεύουν τους ανήλικους χρήστες και ε, όλους ανεξαιρέτως όσον αφορά την ρητορική μίσους και τα μηνύματα που περιέχουν τέτοια ρητορική. Προτείνουμε δηλαδή να τροποποιηθούν ελαφρώς οι ορισμοί έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται και με τα υπόλοιπα μέσα που έχουν προβλεφθεί. Αυτό λοιπόν ε, που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι η πρόταση είναι αρκετά εξισορροπημένη. Φέτος τον Ιανουάριο μας ζητήσατε να ε, δράσουμε ταχύτατα και πιστεύω πως ε, πολύ σωστά κάνατε και μας επιστήσατε την προσοχή στο, στην επίγουσα φύση του θέματος. Τώρα θεωρώ πως όσο πιο γρήγορα έχουμε ένα πλαίσιο τόσο το καλύτερο. Υπάρχει και η ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό. Ε, νομίζω πως έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά προπαρασκευαστικά και εμείς και μαζί με τους ενδιαφερόμενους φορείς και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε σε μία ε, έγκριση χωρίς προβλήματα της πρότασης. Όπω σα είπα, εδώ δεν πρόκειται για την τεχνολογία στην ψηφιακή ενιαία αγορά, αλλά για το τι αυτή σημαίνει για του πολίτε. Και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ε, δείξουμε στου πολίτε ότι μπορούμε να αντιδράσουμε, να αντιδράσουμε γρήγορα και να αντιδράσουμε με τρόπο αποτελεσματικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ε, συνεχίζει να ελπίζει στην ε, συνέχεια αυτή τη πολύ καλή συνεργασία μαζί σα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια πολύ γρήγορη έγκριση τη πρόταση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πράγματι υπήρξε διάλογος αυτή την περίοδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε λοιπόν και τη Γενική σας Διεύθυνση και τον Επίτροπο, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει και κατάλληλο χρονοδιάγραμμα. Εμεί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πρέπει να ε, έχουμε και εμεί το χρόνο μα ε, να εμβαθύνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ λοιπόν για τη σαφήνεια των τριών προτεραιτήτων που μας αναφέρατε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μπόλονς, ε, με την οποία θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα της αξιολόγησης του προγράμματος REFIT και τις ε, ε, επιπτώσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντική η μελέτη επιπτώσεων για μας και θα θέλαμε να μας πείτε τι κάνετε πριν από την πρόταση. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα εξηγήσω και θα σας υπενθυμίσω ποιοι είναι οι αντικειμενικοί στόχοι του εγχείρηματος REFIT που ήταν να πάρουμε την οδηγία και να δούμε εάν το νομοθέτημα αυτό ακόμη εξυπηρετεί τον σκοπό του. Χρειάστηκε δηλαδή να εξετάσουμε εάν οι σκοποί για τους οποίους ψηφίστηκε το νομοθέτημα εξακολουθούν να ισχύουν και αν αντιμετωπίζονται ορθά. Όπως είπε η συναδελφός μου Κλέρ, έπρεπε πρώτα να εξετάσουμε αν υπήρχε λόγος να γίνει απορρίθμιση ή αν υπήρχε λόγος να γίνει ρύθμιση σε άλλους τομείς. Όπως εξήγησε η Κλέρ, βρήκαμε ανάγκη και τα δύο αυτά πράγματα. Όσον αφορά την χώρα προελεύσεως. Ποια ήταν τα αποτελέσματα του REFIT για να καταλήξουν στην πρόταση που εξηγήσαμε. Αυτή η χώρα προελεύσεως είναι καλή υπόθεση. Όπως είπε η Κλέρ, έχει αυξηθεί η διαμεθοριακή διακίνηση. 38% των καναλιών στην Ευρώπη ε, κινούνται διαμεθοριακά. Και για το video on demand, 30% από αυτά που βρίσκεται στην αγορά έρχονται από άλλε χώρε. Άρα ήταν σημαντική πρόοδο και επιτυχία. Και αυτό το refit exercise βρήκε ότι τελικά η αρχή αυτή καμιά φορά στην εφαρμογή της αποδείχνεται περίπλοκη διότι οι κανόνες είναι περίπλοκοι και ιδίω ό,τι αφορά τους μηχανισμούς αποκλήσεων δεν ισχύουν το ίδιο για on demand ή για την linear και γι' αυτό προτείναμε εμεί να αλλάξουμε τους κανόνες. Τώρα, ποια θα είναι η επίπτωση των νέων κανόνων σύμφωνα με την μελέτη αντικτύπου που διαθέτουμε είναι ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους, θα είναι πιο ισότιμοι οι όροι του ανταγωνισμού και on demand και linear και οι καταναλωτές θα ωφεληθούν γιατί πήραμε υπόψη αυτές τις ε, ιδιαιτερότητες των χωρών μελών σε ορισμένες περιστάσεις και όλα αυτά βέβαια οδηγούν σε εξοικονομήσεις και για τους ε, ρυθμιστές και για τις εταιρείες. Σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση, ποια ήταν τα αποτελέσματα του εγχειρήματο REFIT και η ίδια η Κλέα σας εξήγησε ότι έχουν αλλάξει συνήθειες οι θέατες. Η δυνατότητα αλλαγής τώρα switch είναι υψηλότερη και για άλλες μορφές διαφημίσεως όπως τοποθέτηση προϊόντων αλλά και χορηγίες sponsorship δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα ε, είδη διαφημίσεων στην Ευρώπη γιατί οι κανόνες δεν είναι απλοί και γι' αυτό έχει γίνει πρόταση να αλλάξουν. Ποια θα είναι τώρα η επίπτωση της μεγαλύτερης ευελιξίας υπέρ των διαφημιζόμενων. Θα έχουν πιο ισότιμο ε, ανταγωνισμό, άρα μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, περισσότερες επενδύσεις σε διαδικτυακό περιεχόμενο. Θα είναι άσχημο για τους καταναλωτές. Τα αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου είναι ότι υπάρχει βέβαια κάποιο κινδυνο να ενταθούν οι διαφημίσεις στις ε, ώρες αιχμή. Η μελέτη μας όμως δείχνει επίσης ότι υπάρχει και μια... Ε, έχει αλλάξει τόσο πολύ η ελαστικότητα της ζήτησης που συνήθως οι broadcaster προβαίνουν σε αυτοπεριορισμό για να μην χάσουν θεατές. Νομίζουμε λοιπόν ότι δεν θα υποστεί μια ο καταναλωτή και εν πάση περιπτώσει εάν σε μια συγκεκριμένη χώρα μέλος φανεί ότι η αγορά δεν ακολουθεί όπως δεν ε, εξελίσσεται όπως είπαμε, μπορούμε πάλι να αλλάξουμε τους κανόνες. Για, τη, για τους κανόνες προστασίας των ανηλίκων. Το REFIT βρήκε ότι ρυθμίζουμε την τηλεόραση, ενώ αυτά που κάνουν τα παιδιά είναι να παρακολουθούν on demand, video on demand. Άρα οι κανόνες δεν παρακολουθούσαν την πραγματικότητα. Οι περισσότερες δε χώρες μέλη έχουν εφαρμόσει αυστηρότερους κανόνες στον τομέα αυτό. Και γι' αυτό, όπως είπε η Κλέρ, προτείναμε να εφαρμόζονται ακριβώς οι ίδιοι κανόνες. Τώρα, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των νέων κανόνων, βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών, των ανηλίκων, μεγαλύτερη εναρμόνιση, γιατί οι περισσότερες χώρες μέλη εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες, τώρα θα πρέπει όλες να εφαρμόζουν τους αυστηρότερου κανόνες. Αυτό θα σημάνει και υψηλότερο κόστος για τον κλάδο. Καταρχήν ναι, αλλά υπάρχουν ήδη κανόνε, δηλαδή δεν αρχίζουμε από το μηδέν και βέβαια και οι περισσότερες χωρισμένοι μέλη τους εφήρμοζαν ήδη για την προβολή ευρωπαϊκών έργων. Τα αποτελέσματα πάλι του Ρεφίτ ήταν ότι υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός. Οι υφιστάμενοι κανόνες για την προβολή των ευρωπαϊκών έργων on demand δεν έχουν επιφέρει καμιά εναρμόνιση είναι τόσο ανοιχτοί και τόσο ασαφείς οι κανόνες που οι χώρες μέλη έχουν πάρει πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις κάτι το οποίο οδήγησε σε έλλειψη ίσων όρων ανταγωνισμού και μέσα στις ίδιες τις χώρες μέλη ανάμεσα στους διάφορους φορείς. Ήταν λοιπόν καθαρό ότι κάτι έπρεπε να γίνει. Αυτό έχει επιπτώσεις και στο επίπεδο επενδύσεων, διότι αν συγκρίνουμε το επίπεδο επενδύσεων σε ευρωπαϊκά έργα από τους broadcaster και από τους φορείς του video on demand είναι πολύ διαφορετικά. Μιλούμε για 20% και λιγότερο από 1% για το video on demand. Και γι' αυτό προτείναμε να αλλάξουν οι κανόνες, όπως αναφέρθηκε ήδη. Και ποια θα είναι η επίπτωση των νέων κανόνων, σύμφωνα πάλι με τη μελέτη αντικτύπου μας, θα, είναι βέβαια, θα ωφεληθεί βέβαια γενικότερα το πολιτιστικό γίγνεσθε. Θα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση οι πολίτες σε ευρωπαϊκά έργα, θα είναι καλύτερα για την ισότητα ανταγωνισμού, διότι τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα όσα κάνει broadcaster και το on demand, θα σημάνει κάποιο κόστος για τον κλάδο και για τους ε, video on demand players. Ναι, όχι όμως τόσο πολύ, διότι η ανάλυση μας μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σύστημα για βίντεο on demand βασίζεται σε ένα σύστημα revenue sharing, δηλαδή ε, διαμοιρασμού των ε, ε, εσόδων. Από την άλλη μεριά, αυτό που προτείνουμε είναι να ληφθεί υπόψη το μέγεθος των ε, εταιριών. Προβλέπουμε λοιπόν μια υποχρεωτική εξαίρεση υπέρ των μικρών επιχειρήσεων για να ληφθεί υπόψη αυτή η έξτρα αύξηση κόστους. Αυτά για την προβολή των ευρωπαϊκών έργων. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πλατφόρμες, ποια ήταν τα αποτελέσματα του εγχειρήματο Refit. Ο στόχο για την προστασία των ανηλίκων και των πολιτών από κηρύγματα μίσους εξακολουθεί να ισχύει, δεν έχει επιτευχθεί ωστόσο, διότι στον ε, επιγραμμικό κόσμο δεν υπάρχουν κανόνες. Αν δείτε τι κοιτάζουν οι ανήλικοι, θα δείτε σε πολλές ε, χώρες ε, παρακολουθούν περισσότερο διαδικτυακό περιεχόμενο παρά τηλεόραση. Και οι μελέτες μας έδειξαν μάλιστα ότι οι ανήλικοι ταυτίζουν ορισμένες, ορισμένους δικτυακούς τόπους με ε, πορνογραφία και βία. Γι' αυτό προτείναμε εμείς εν τέλει να επεκταθεί η ισχύ των κανόνων για να ληφθούν υπόψη αυτές οι δύο ανησυχίες. Ποια, ποιες θα είναι οι συνέπειες των νέων κανόνων, ε, καλύτερη προστασία των ανηλίκων και των πολιτών απέναντι σε κηρύγματα μίσους θα είναι καλό και για την ενιαία αγορά, διότι βρισκόμαστε πάντοτε μέσα στο χρονικό πλαίσιο, δηλαδή προλαμβάνουμε τον κατακαιρματισμό. Οι χώρες μέλη μπορούν να κατευθυνθούν σε πολλές κατευθύνσεις. Σε ένα τομέα όπου γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πλατφόρμες που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχει λοιπόν επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το πεδίο του ανταγωνισμού, διότι άλλοι υφίστανται τις ρυθμίσεις, άλλοι φορείς όχι, θα υπάρξει, θα σημάνει αυτό κάποιο κόστος για τις πλατφόρμες. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι ήδη πολλά γίνονται. Υπάρχει πολύ λοιπόν αυτορύθμιση. Πάλι λοιπόν δεν αρχίζουν από το μηδέν όλοι αυτοί. Μέχρι τώρα λοιπόν τα αποτελέσματα που δείχνει ε, το εγχείρημα REFIT είναι ότι υπάρχει ανάγκη για αλλαγές και αυτά που προτείνουμε θεωρούμε ότι είναι ισορροπημένα. Ορίστε κυρία Πρόεδρε, αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανάλυση. Συνοπτική μεν, αλλά πολύ σαφής ε, επί των θεμάτων αυτών. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο έχετε τροποποιήσει και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, το θέμα των ρυθμιστών. Μεγαλύτερη ανεξαρτησία λοιπόν και ε, μεγαλύτερος ρόλος ε, των ρυθμιστών σε θέματα συντονισμού, ε, διότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι και η αποτελεσματικότητα των του σεβασμού αυτών των κανόνων. Ε, υπάρχουν ε, στις χώρες μας προβλήματα, ε, κυρίως σε θέματα προστασίας των ανηλίκων, που δεν καλύπτονται πάντα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να δώσουμε πρώτα το λόγο στις δύο συνεισηγήτριες. Η κυρία Πρώτα ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έλαβε τον κόπο να έλθει και να μας εξηγήσει το σχέδιο για να αρχίσουν και συζητήσει στην Επιτροπή Πολιτισμού. Είναι σωστή η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προτίμησε μια εξέλιξη και όχι μια επανάσταση, διότι έχουμε νέες τεχνολογίες, έχουμε νέους τρόπους μεταδόσεων αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και οι παλαιοί τρόποι μεταδόσεως που καμιά φορά μάλιστα κερδίζουν έδαφος. Αναμέσων όρο βλέπουν οι άνθρωποι τέσσερις ώρες τηλεόραση την ημέρα. Δεν μπορεί λοιπόν να πει κανείς ότι πεθαίνει η παραδοσιακή τηλεόραση. Ίσως οι εξελίξεις να αλλάξουν στο μέλλον, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται, χρειάζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού και για τα δύο είδη τηλεοπτικών υπηρεσιών και on demand και τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο. Είναι σωστή λοιπόν η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως είπα στο σημείο αυτό. Είναι σωστό επίσης να υπάρξει μια ευκαμψία στο θέμα των διαφημίσεων ανάμεσα στο linear και στο non-linear που τώρα μέσα στο τεχνικό περιβάλλον που διαθέτουμε δεν είναι πλέον δυνατός αυτός ο διαχωρισμός. Διότι ακόμα και στο linear, στη γραμμική δηλαδή μετάδοση, συνήθως το μηχάνημά μου έχει και ένα σκληρό δίσκο, ακόμα και αν διακόψω λοιπόν την ε, παρακολούθηση, μπορεί να συνεχίσει να γράφεται η εκπομπή και μετά να το παρακολουθήσω αργότερα. Λόγω λοιπόν των τεχνικών δυνατοτήτων που ανοίγονται τώρα πλέον, κάποια στιγμή και η γραμμική μετάδοση θα γίνει μη γραμμική. Πολύ σωστά λοιπόν προχωρείται σε μια μεγαλύτερη ευκαμψία η ευελιξία. Για τις υπηρεσίες on demand βρίσκω σημαντικό, πολύ σημαντικό, να προστατευτούν περισσότερο οι ανήλικοι, διότι όλο και περισσότερο νέα παιδιά και ανήλικοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Video On Demand. Για τη συζήτηση που έχει αρχίσει ήδη, ε, αν δει κανείς τους τίτλους των εφημερίδων και των ειδικών περιοδικών για την προβολή ευρωπαϊκών έργων, εγώ βρίσκω ότι κάνουμε καλά και κάνουμε το βήμα αυτό για να προωθηθούν ευρωπαϊκά έργα και στις διάφορες πλατφόρμες. Υπάρχουν πλατφόρμες που έχουν κάνει από μόνες τους το βήμα αυτό. Μεγάλες πλατφόρμες οι οποίες έχουν και ένα τμήμα ευρωπαϊκής παραγωγής. Αν θέλει όμως κανείς να βρει απήχηση στο κοινό, θα πρέπει να προβάλλει και ευρωπαϊκές παραγωγές διότι η οπτικοακουστική αγορά μας εξακολουθεί να διέπεται από την πολιτιστική πολυφωνία που διαθέτουμε στην Ευρώπη. Και είναι σημαντικό λοιπόν να έχει υπόψη του κανείς ότι η κάθε Ιταλική τηλεοπτική σειρά δεν ε, ενδιαφέρει πάντα απαραίτητα και τους Γερμανούς τηλεθεατές. Κάθε ε, Βρετανική αστυνομική σειρά μπορεί να μην ενθουσιάζει τους Ιταλούς. Δεν χρειάζεται λοιπόν να γίνει αυτή η ε, από το πίσω παράθυρο προσπάθεια εξίσωσης της ε, πολιτιστικής παράδοσης στην Ευρώπη. Για τις ε, υπηρεσίες on demand βρίσκω σωστό επίσης να συμμετέχουμε και στη δημιουργία διαδικτικού περιεχομένου είτε μέσω των ταμείων είτε μέσω και ιδίων παραγωγών που θα συμβάλλουν ευρωπαϊκές ίδιες παραγωγές. Το αν θα αναγνωριστούν ότι έχουν κάποια αξία ή όχι, αυτό θα το δούμε. Και θα πρέπει να συζητήσουμε το μοντέλο που θα ακολουθήσουμε. Πολλά θα τα αναλάβουν οι χώρες μέλη. Και είναι αλήθεια ότι οι χώρες μέλη διαθέτουν μεγάλο περιθώριο ελιγμών και αποφάσεων για το πώς θα προωθήσουν τις ευρωπαϊκές παραγωγές και αν θα συμμετάσχουν και με ποιο τρόπο για τις πλατφόρμες video sharing για μένα είναι σημαντικό πάλι εδώ να τονιστεί η προστασία των νέων γιατί και οι ευθύνε σημαντικές είτε πρόκειται για το YouTube ή άλλα σχετικά κανάλια και άλλες πλατφόρμες πρέπει να προβλεφθεί προστασία των ανήλικων και να είναι εξασφαλισμένη διότι είναι τέτοια η επιρροή στον ψυχισμό των νέων των ε, πλατφορμών αυτών πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη αυτά. Πρέπει να αντιμετωπιστούν λοιπόν σωστά οι ανάγκες των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας μας. Και για τα κηρύγματα μίσους ακριβώς το ίδιο ισχύει. Γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει περιλάβει και το θέμα αυτό και με σωστό τρόπο. Ένα θέμα ακόμη ωστόσο, έρχομαι στο τελευταίο, το ζήτημα της accessibility. Εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού έχουμε συζητήσει και για το Accessibility Act ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των διαφόρων κανονισμών. Και δεν είναι σωστό αυτό. Εγώ θα ήθελα να έχει να παίξει μεγαλύτερο ρόλο η accessibility στον κανονισμό και να μην υπάρξει μονάχα το ξεχωριστό accessibility act. Χρειάζεται ειδικό ορισμός διότι εάν βάλουμε, αν επιβάλλουμε μια συνολική υποχρέωση σε όλα τα οπτικοακουστικά περιεχόμενα που υπάρχουν παντού για την accessibility, για την προσβασιμότητα δηλαδή, ε, υπάρχουν και προϊόντα πολύ εξειδικευμένα για πολύ εξειδικευμένο κοινό. Να μην μειωθεί η ποικιλία των ε, προϊόντων και των παραγωγών. Τάσομαι υπέρ μιας ε, πιο ξεκάθαρης υποχρέωσης των παρόχων να εξασφαλίζουν αυτήν την accessibility, την προσβασιμότητα ώστε η κοινωνία ολόκληρη να μπορεί να συμμετέχει. Αλλά θα πρέπει να χρειαστεί να, μάλλον θα χρειαστεί να το εξετάσουμε εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού και να τα βγάλουμε αυτά τα πράγματα από το Accessibility Act. Ευχαριστώ πολύ. Η Πέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σήμερα προσπάθησε να μας παρουσιάσει την πρότασή της και να μας ενημερώσει και μάλιστα εν ώψη της εκτιμήσης αντικτύπου που έχει γίνει. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες θετικές πτυχές τις οποίες μπορώ να αναγνωρίσω στην πρόταση. Υπάρχουν όμως και κάποια σημεία για τα οποία θα ήθελα περισσότερες ε, λεπτομέρειες και δεν με ευχαριστούν τόσο. Ε, καλωσορίζω βέβαια τα θετικά στοιχεία, δηλαδή τις ρυθμίσεις για τη χώρα προέλευσης. Πιστεύω πως η απόφαση ήταν πολύ σωστή και ε, μας οδήγησε σε μια διεύρυνση της ε, αγοράς, γι αυτό, λοιπόν, ψηφιακής αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως αυτή η αρχή είναι πολύ καλό που διατηρείται. Ε, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ε, διευκρινήσεις που χρειάζονται ιδιαίτερα για τις εξαιρέσεις και τις ιδιαιτερότητες των κρατών ε, μελών. Γι' αυτό λοιπόν θα επιθυμούσα να είναι λίγο πιο σαφής η διατύπωση από ό,τι τώρα. Σε γενικές γραμμές όμως νομίζω πως είναι πολύ σωστό να διατηρηθεί αυτή η αρχή τώρα. Η τελευταία αναθεώρηση τη ε, οδηγία για τα οπτικο-ακουστικά μέσα έγινε πριν από 7 χρόνια. Αυτό μας δείχνει πόσο γρήγορο έχει γίνει ο κόσμος μας, ιδιαίτερα στο νοπτικό ακουστικό ε, χώρο. Και αυτό λοιπόν θεωρώ πως ε, τώρα Χρειαζόμαστε μια νομοθεσία η οποία θα μας εξασφαλίσει με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, έτσι ώστε ε, να μπορούμε να προβλέψουμε καταστάσεις. Σίγουρα δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο κόσμος σε 10 χρόνια, όμως γι' αυτό πιστεύω πως χρειάζεται ε, μια οδηγία η οποία δεν θα χρειαστεί να αναθεωρηθεί μετά από 6-7 χρόνια. Πρέπει να είμαστε ένα βήμα πέρα από τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Γι' αυτό θεωρώ πως θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε εάν θα μπορούσε να, αν θα μπορούσαμε να αλλάξουμε κάπως την ε, διατύπωση σχετικά με τις γραμμικές και τις ε, επιγραμμικές συνδέσεις. Η Σαμπίνα Φερχάιεν ήδη μας είπε ότι για τους πολίτες δεν έχει καμία απολύτως σημασία το, ότι, ε, το, το αν το περιεχόμενο που καταναλώνουν είναι επιγραμμικό ή γραμμικό. Αυτή τη στιγμή όταν κάποιος έχει ένα κινητό δεν μπορεί να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στην τυπική κλασική τηλεόραση ή σε μια υπηρεσία on demand. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως έτσι όπως αλλάζουν τα πράγματα πρέπει εμείς εδώ να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτές ε, τις ε, διαφορές. Τώρα. Θεωρώ πως και αυτή η δυνατότητα περισσότερης ευελιξίας για τις διαφημίσεις είναι κάτι καλό. Είναι κάτι που ζητούσαμε εξάλλου από αρκετό καιρό και πιστεύω πως ε, θα πρέπει οι παραδοσιακοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς να αναλογιστούν πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτήν τη νέα ευελιξία πώς θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν. Διότι αν δεν τη χρησιμοποιήσουν με σωστό τρόπο, τότε θα ε, χάσουν τηλεθεατές, θα χάσουν ακροατές και θα χάσουν κατά συνέπεια εισόδημα και από τις διαφημίσεις. Πολλές φορές ε, όταν γίνεται λάθος χρήση ε, των διαφημίσεων ε, παρατηρείται ότι ο τηλεθεατής αλλάζει κανάλι, δεν θέλει να δει διαφημίσεις. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως εδώ μπορώ να πω και χαίρομαι που το λέω και ως δημοκράτης ότι έχουμε μία πρόταση η οποία φροντίζει προς, ε, φροντίζει τους πολίτες, διότι αν ο τηλεθεατής είναι δυσαρεστημένος τότε θα αλλάξει κανάλι. Πιστεύω πως είναι σωστή λοιπόν η προσέγγιση. Ωστόσο, στις διαφημίσεις υπάρχει ένα σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο τι επιτρέπεται σε, γραμμικές, ε, σε γραμμικό περιεχόμενο και τι σε μη γραμμικό περιεχόμενο, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των ε, ανηλίκων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαφημίσεις που προορίζονται για παιδιά και θα μπορούσαμε ίσως εδώ να δούμε το κείμενο και να δούμε εάν χρειάζεται κάποια πρόσθετη ρύθμιση για το γραμμικό περιεχόμενο και για το επιγραμμικό online. Ίσως θα μπορούσε να γίνει κάποια πρόβλεψη για ε, συνομοθέτηση ή για ε, αυτορύθμιση. Να δούμε αν θα είναι κάτι το οποίο θα ελέγχεται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή θα υπάρχει κάποιο αμοιβαίο σύστημα ελέγχου που θα συμμετέχουν και οι πάροχοι. Τώρα θεωρώ πως στο μέλλον θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο το θέμα της ε, δημοσιογραφικής ε, ευθύνης. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία απολύτως διαφορά επιγραμμικά ή γραμμικά. Αλλά πρέπει να δούμε, πιστεύω, πού υπάρχει η ευθύνη των ε, δημοσιογράφων, η ευθύνη των συντακτών και ίσως χρειάζεται διαφορετική ε, νομοθεσία για αυτήν την περίπτωση παρά για το γενικότερο περιεχόμενο και για το generated content. Επίσης εδώ είναι και πολύ σημαντικό να δούμε την ε, πολυμορφία απόψεων. Εδώ πιστεύω πως έχει γίνει ένα βήμα προς την ε, επιθυμητή κατεύθυνση και για τις πλατφόρμες video sharing. Πιστεύω πως έχουν γίνει αρκετά, ωστόσο ε, πρέπει να δούμε πως ε, πρέπει να δούμε ότι χρειάζεται να διατηρηθεί η ευθύνη του περιεχομένου και να ε, φροντίσουμε να μην απομακρυνθούμε πολύ από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Χρειάζεται δηλαδή μία αστυνόμευση τροποντινά του διαδικτύου, έτσι ώστε να αποφεύγονται ε, παρανομίες, να αποφεύγεται ρητορική μίσους, να προστατεύονται οι ανήλικοι χρήστες. Γι' αυτό χρειάζεται όταν ε, διαπιστώνονται τέτοιες παραβιάσεις να λαμβάνονται μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν εδώ η αρχή της, ε, του αυτοέλεγχου, της αυτορύθμισης πιστεύω πως πρέπει να διατηρηθεί και να αναπτύξουμε διάφορα τέτοια συστήματα, αλλά και συστήματα συνεργασίας στον έλεγχο του περιεχομένου. Και ας μην διστάσουμε λοιπόν να είμαστε ε, προορατικοί γι' αυτό. Τώρα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να λάβει υπόψη και την απόφαση του δικαστηρίου για τα ε, ενσωματωμένα βίντεο τα βίντεο δηλαδή τα οποία είναι ενσωματωμένα σε ένα άρθρο δεν υπόκειται στην οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα. Υπάρχουν όμως ε, κατηγορίες βίντεο. Κάποια βίντεο τα οποία ας πούμε είναι ενσωματωμένα σε, μια, σε έναν ιστότοπο εφημερίδας τότε πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία. Πιστεύω πως αυτή είναι μια σωστή προσέγγιση και έχετε κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και προς το να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού ανάμεσα στους ε, παρόχους ε, ειδησιογραφικού περιεχομένου, τους παραδοσιακούς και τους ε, νεότερους. Τώρα, πρέπει να πω πως δεν αγαπώ τους ποσοστώσεις καθόλου και πιστεύω πως αυτό είναι μια πατερίτσα για να στηρίξουμε τα ευρωπαϊκά έργα. Όμως, τίνω εδώ να προτιμώ μία ίση μεταχείριση ανάμεσα στο γραμμικό και στο μη γραμμικό περιεχόμενο. Γραμμικό περιεχόμενο λοιπόν έχουμε μια ποσόστοση του 30%, επιγραμμικό 20%. Ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε αυτά τα ποσοστά για να δούμε αν μπορούμε να ε, τα εξισορροπήσουμε και να δούμε πώς μπορούν αυτές οι πλατφόρμες βίντεο να, να ε, έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση από τα ταμεία, έτσι ώστε να δημιουργούν ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Θεωρώ πως θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε, θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και τις πλατφόρμες βίντεο sharing στη, σε, αυτό, σε αυτά τα ταμεία και την πρόσβαση του στη χρηματοδότηση. Τώρα, συνδεδεμένη τηλεόραση, Connected TV. Υπάρχει μία έκθεση πρωτοβουλίας σχετική. Για μένα αυτά, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ σημαντικό να δίνουν την δυνατότητα στις αιτιολογικές σκέψεις να μεταφερθούν η διατάξη για την ασφάλεια δικαίου στα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να τους δοθεί αυτή η δυνατότητα, προσβασιμότητα. Η Σαμπίνα Φερχάη νομίζω τα είπε όλα. Υπάρχει μια σχετική πρόταση από εμένα για την προσβασιμότητα, για το Accessibility Act. Εδώ χρειάζονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις και πρέπει οι ρυθμίσεις αυτές να βρίσκονται αγκυροβολημένες στην οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα. Θεωρώ όμως ότι θα είμαστε πιο γρήγοροι ε, με την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα παρά με την ε, οδηγία για την προσβασιμότητα. Εξαρτάται βέβαια και από το Συμβούλιο, αλλά σίγουρα ε, νομίζω πως πρέπει να διασφαλιστεί και στις δύο περιπτώσεις η διαφάνεια και ελπίζω να είμαστε γρήγοροι, να εργαστούμε με γρήγορους ρυθμούς έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε σύντομα και η διαφάνεια να είναι κύριο μέλημά μας. Θα συζητηθεί και όλας ελπίζω στην ε, συνάντηση με τους ε, διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. Ελπίζω λοιπόν να συνεισέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χέλικα Τρούπελ τώρα. Θα ήθελα να ζητήσω από τους σκιώδεις ε, την κυρία Τρούπελ, τον κύριο Τόμ, δεν ξέρω ποιος άλλος θέλει να παρέμβει, η κυρία Τιλόλφη, την άλλη συνάδελφο δεν τη βλέπω, θα ήθελα να δω ποιοι θέλουν το λόγο. Ωραία. Ξεκινάμε με την κυρία Τρούπελ. Τέσσερα λεπτά ο καθένας παρακαλώ για τους και Ευχαριστώ και από τη δική μου πλευρά τις ε, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και της κυρίας Χάιεν και Κάμερ Εβερτ. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής στα οπτικοακουστικά είναι σωστή και σημαντική, διότι η τεχνολογική εξέλιξη το απαιτεί, να προσαρμοστούν δηλαδή οι ρυθμίσεις. Και γι' αυτό είναι σημαντικό οι τρεις μεγάλοι τομείς, είτε πρόκειται για γραμμική τηλεόραση, τηλεόραση είτε για video on demand, είτε για video sharing, είναι σημαντικό να περιληφθούν. Επίσης, προστασία των ανηλίκων, προστασία κατά των κηρυγμάτων μίσους. Πρέπει να υπάρχουν αυστηροί κανόνες και για το video on demand και τι πλατφόρμες video sharing. <clears throat> για το ερώτημα τώρα τη προβολής ευρωπαϊκών έργων, ευρωπαϊκών παραγωγών. Και εκεί είναι σημαντικό να υποχρεωθούν οι πλατφόρμες video on demand να προσφέρουν τουλάχιστον 20% ευρωπαϊκών έργων. Υπάρχει και το αντεπιχείρημα ότι έτσι θα γίνουν λιγότερο ελκυστικές ή ότι θα αφαιρέσουν άλλες προσφορές έργων. Εγώ δεν νομίζω. Εγώ θεωρώ ότι οι ευρωπαϊκές αγορές είναι όντως έτσι που πρέπει να προσφέρονται και ευρωπαϊκές παραγωγές γιατί αλλιώς δεν είναι ελκυστικές πλέον οι πλατφόρμες αυτές για τους θεατές, για τους καταναλωτές, για την ε, συμμετοχή σε χρηματοδότηση ευρωπαϊκών παραγωγών επίσης είμαι σύμφωνη. Το θέμα είναι τώρα επίσης της δυνατότητας προσβασιμότητας στις διάφορες, τις ε, διάφορες αυτές παραγωγές. Η δυνατότητα ανείχνευσής τους δηλαδή στις διάφορες πλατφόρμες. Αυτό πρέπει επίσης να περιληφθεί όχι μόνο στα εκτιμώντα, αλλά και στο ίδιο το νομοθετικό κείμενο. Και η αρχή της χώρας προελεύσεως πρέπει να παραμείνει ενισχύ, γιατί είναι από τις βασικές αρχές λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Τώρα, για την ρύθμιση των ε, διαφημίσεων πρέπει να υπάρχει πάντοτε ξεκάθαρη διάκριση, ξεκάθαρος διαχωρισμός ανάμεσα στο κατά αυτό περιεχόμενο και στην διαφήμιση. Γι' αυτό και δεν μου αρέσει αυτό το product placement, να επιτραπεί δηλαδή η έμεση τοποθέτηση προϊόντων. Έτσι δεν θα μπορέσω να συμφωνήσω σε αυτό. Επίσης δεν είμαι και υπέρ αυτή τη διακοπή των εκπομπών ανά 20 λεπτά για να προβληθούν διαφημίσεις. Σωστό μου φαίνεται, ότι, ε, σωστό μου φαίνεται να πούμε ότι υπάρχει κάποια ευκαμψία ή κάποια ευελιξία, δηλαδή η διαφήμιση να κατανέμεται σε ολόκληρη την ημέρα και να μην υπολογίζεται αναώρα εκπομπής. Κάτι που θέλω να διασφαλιστεί είναι η ακυρότητα του σήματος. Έχουμε το φαινόμενο ότι η διαφήμιση πέφτει πάνω στα μηνύματα, ειδήσει κλπ. χωρίς να ρωτούν τους διαμορφωτές των εκπομπών. Αυτό θα πρέπει να γίνει μονάχα με την έγκριση του υπευθύνου του προγράμματος. Αυτό δεν ρυθμίζεται επαρκώς στην ε, ε, πρόταση. Σωστό είναι επίσης να υπάρχει ένα όργανο των ανεξάρτητων ρυθμιστών και αυτοί να έχουν και την υποχρέωση σχετικά για την παρακολούθηση των μηνυμάτων που ευθύνονται σε νέους καθώς και των κηρυγμάτων μίσους. Ακούμε συχνά, μάλλον θα πρέπει να μαθαίνουμε συχνά πώς ρυθμίζουν τα πράγματα αυτά και αν όντως ρυθμίζουμε τον τρόπο που αναμένουμε. Για την πρόσβαση ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες. Και εκεί νομίζω ότι καταρχήν μέσα στην οδηγία για τα οπτικοακουστικά θα πρέπει να περιληφθεί και η σχετική μνήμα. Όλοι ενδιαφέρονται ώστε τα προγράμματα είναι έτσι φτιαγμένα που άνθρωποι με διάφορες αναπηρίες να έχουν καλύτερη προσβασιμότητα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια σύγκρουση στόχων σε ό,τι αφορά την προσφορά πολιτιστικής πολυφωνίας. Όμως θεωρώ ότι πρέπει να, υπάρξουν να υπάρξει μεγαλύτερη προσφορά περιεχομένου που να απευθύνεται και σε ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες. Και μια παρατήρηση τώρα για την ευθύνη που προέρχεται από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει να σκεφτεί κανείς όμως αν θα πρέπει και να υπάρξει κάποια διευκρίνηση. Εκεί δηλαδή όπου γίνεται σύσταση για κάποιο περιεχόμενο και δεν πρόκειται απλώς για αναμετάδοση, αλλά όπου ένας πάροχος κάνει ίδια προσφορά και με τον τρόπο αυτό αποκτά ιδιαίτερη ελκυστικότητα και επομένως διαφημίσεις, πρέπει να δούμε πώς έχει ρυθμιστεί εκεί στην οδηγία ηλεκτρονικού εμπορίου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έρεται η ευθύνη. Αλλά χρειάζεται μια διευκρίνηση για να υπάρξει και μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Εν τέλει, όταν τίθεται το ερώτημα, Ποια είναι η ευθύνη και μέσα σε αυτήν βάζω και τον αυτοπεριορισμό των παρόχων ε, διαδικτυακού περιεχομένου. Ευχαριστούμε τη Χέλντα. Για να περάσουμε στους άλλους και οδησίγητες, η κυρία Τόμ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις δύο συνεισηγήτριες για την προσπάθεια και το χρόνο που έχουν αφιερώσει και θα εκφράσω κάποιες από τις θέσεις της ομάδας. Ε, βάσει των ε, πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων ε, πρέπει να αναθεωρήσουμε την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, επομένως είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις για να εξυγχρονίσουμε την πρόταση. Θα αναφέρω δύο εξ αυτών, διότι είναι αρκετά εκτεταμένη η πρόταση. Πρώτον, η πρόταση απλουστεύει τους κανόνες βάσει των οποίων καθορίζεται ποιο κράτος μέλος έχει τη δικαιοδοσία, τη λεγόμενη αρχή της χώρας προέλευσης. Ξέρετε ότι αυτό είναι θέμα διαμάχης μεταξύ κρατών μελών. Δεύτερον, η πρόταση επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και επομένως εφαρμόζεται και για πλατφόρμες ανταλλαγής ε, βίντεο περιεχομένου. Επομένως ε, υπάρχουν κατάλληλε διατάξει για πλατφόρμες ανταλλαγή περιεχομένου βάσει συγκεκριμένων προποθέσεων. Ο ορισμός βέβαια έχει κάποια προβλήματα, κυρίως στην πρακτική του εφαρμογή. Θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά πού βρίσκονται τα όρια του ορισμού και σε ποιο βαθμό θα υπάρχει διαφορετική ε, μεταχείριση των διαφόρων ε, ε, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της, των, της πλατφόρμας που διαθέτει το καθένα. Η οδηγία αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απομακρύνεται ε, από την παραδοσιακή τηλεόραση ως ε, το σημείο αναφοράς. Επίσης έχουμε την ε, απαγόρευση της ρητορικής μίσους που όπως ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί από την παρούσα απόφαση πλαίσιο για την έκφραση κάποιων μορφών μίσους, ρατσισμού και ξενοφοβίας ευπρόσδεκτη μεν η πρόταση, αλλά υπάρχουν κάποιες πρακτικές ε, δυσκολίες στην εφαρμογή της. Πώς θα επηρεάσει την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για παράδειγμα, που προστατεύει τις διαδικτυακές πλατφόρμες από την ευθύνη για το ε, περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες. Επίσης, ε, τι γίνεται και πώς μπορούμε να παρακολουθούμε τους χρήστες και κυρίως πώς θα απομακρύνουμε τις σχετικές απειλές για τους χρήστες. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν προσεκτικά τα διάφορα στοιχεία της οδηγίας και θα πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία. Θα πρέπει βεβαίως ε, να ε, ε, προσέξουμε γιατί μας περιμένει πολλή δουλειά. Δεν ήθελα εδώ βέβαια να μιλήσω για 5 ή 10 ή 15 λεπτά, αλλά αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που θα συζητήσουμε το ζήτημα και έχω 12 ερωτήσεις. Σήμερα ανέφερα μόνο τις δύο εξ αυτών. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντινόλφη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου με μια γενική παρατήρηση, στην οποία αναφερθήκατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά τη θέση των δύο συγητών για τον κώδικα δεοντολογίας. Ε, μου το επιβάλλει ε, η πειθαρχία και η τιμή με την οποία προσπαθώ να ασκήσω τα καθήκοντά μου. Ε, θα πρέπει να έχουμε ένα ε, στοιχείο, ένα νομοθέτημα το οποίο δεν θα πρέπει να στερείται ηθικής και διοντολογίας. Υπάρχει το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων για τις δύο συνεισηγήτριες και ελοχεύει ο κίνδυνος να υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα σύγκρουσης συμφερόντων. Πρέπει να γίνει μια δημόσια συζήτηση και διάφανη συζήτηση όπως αυτή που κάναμε χθε στους συντονιστές και πρέπει το Κοινοβούλιο να εξετάσει την υπόθεση και να επιλύσει το πρόβλημα διαπαντός. Αλλιώς θα ε, επικρέμεται από πάνω μας ως δαμάκλειος ε, σπάθη και μπορεί και οι πολίτες να μας κατηγορήσουν ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι και δεν είμαστε υπεράνω πάση υποψίας. Εγώ δεν θα ήθελα να επαναλευθούν οι σκηνέ που είδαμε στην Ιταλία με τον πρώην Πρωθυπουργό Μπερλουσκόνη. Και μάλιστα μας έχει μάθει και κάτι ο κύριος Μπερλουσκόνη. Οι πιθανές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει να επιλύονται αμέσως. Αλλιώς ελοχεύει ο κίνδυνος να ε, διαιωνίζεται η κατάσταση και φυσικά να ε, αμαυρώνεται η φήμη και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των ε, ίδιων των ευρωβουλευτών και να μην μπορούμε να ασκήσουμε σημαντικά το έργο μας. Θα πρέπει λοιπόν να ε, θέσουμε το θέμα στον πρόεδρο Σούλς και στη Συμβουλευτική Επιτροπή για να επιληθεί μια για πάντα το θέμα. Τώρα, όσον αφορά την οδηγία, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία εντάχει. Καταρχάς, η διά, ε, ε, γραφή της διάκρισης μεταξύ γραμμικών και μη γραμμικών υπηρεσιών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, διότι υπάρχουν κάποιες φαιές ζώνες, τις οποίες είναι ακόμα χρήσιμη αυτή η διάκριση. Και κατά την άποψή μου θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο καλύτερα το ζήτημα και να δούμε κατά πόσον πρέπει να διαγράψουμε αυτή τη διάκριση ή όχι. Δεύτερη παρατήρηση, αρχή της χώρας προέλευσης. Ναι, μεν η αρχή αυτή ήταν ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα παρέχονται οι υπηρεσίε μια άλλη χώρα, αλλά θα πρέπει να είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο προ μια ενιαία αγορά ένα ενδιάμεσο στάδιο μιας ψηφιακής ενίας αγοράς χωρίς γεωγραφικούς φραγμούς, χωρίς τεχνικούς ε, κατακαιρματισμούς της αγορές. Επομένως αυτή είναι η δέσμευσή μας. Τρίτον, σύστημα ποσοστώσεων προαγωγής ευρωπαϊκών έργων. Σίγουρα είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό μεν, αλλά προς το παρόν έχει αποδείξει ότι δεν έχει αποτέλεσμα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στην Ιταλία με την Agicom για παρεκκλήσεις για την Disney και τη Mediaset. Επομένως πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα ε, πλαίσια τα οποία θα προστατεύουν τα ευρωπαϊκά έργα με αυτόνομο τρόπο. Τέταρτον, προστασία των ανηλίκων και διαφήμιση. Στην Ιταλία ο συνάδελφος Ρομπέρτο Φέκο κέρδισε μια μάχη ε, και κατάφερε να μην μεταδίδεται διαφήμιση σε ένα δημόσιο ε, κανάλι για παιδιά, το, στο Ιραϊούνα και ζήτησε να καταργηθεί η διαφήμιση σε όλα τα κανάλια τα οποία προσφέρουν παιδικό περιεχόμενο και είναι για παιδιά. Ε, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε την ίδια άγουσα και στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφήμιση σε κανάλια τα οποία είναι της δημόσιας τηλεόρασης. Εγώ δεν είμαι σε καμία περίπτωση υπέρ του ε, ποσοστού της διαφήμισης και άλλωστε και η εμπορική τηλεόραση αν θέλει να επιβιώσει θα πρέπει να είναι σε θέση να ε, ε, εξυγχρονιστεί. Πέμπτη πτυχή. Ανεξαρτησία όσων καλούνται να εποπτεύουν τη ραδιοτηλεοπτική αγορά. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες για τους φορείς που πρέπει να εποπτεύουν την αγορά και θα πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητοι. Όσοι είναι ε, φορείς εποπτείας της αγορές θα πρέπει να μην έχουν καμία πολιτική εξουσία. Εδώ δίδαγμα Μπερλουσκόνη και πάλι θα μπορούσε να υπάρχει ένα σύστημα χρηματοδότησης αυτών των αρχών, θα μπορούσε να προβλέπεται τμήμα των εσόδων που έρχονται από την κατανομή των συχνοτήτων να δίνονται στις ανεξάρτητες αυτές αρχές, ώστε να υπάρχει αυτόνομη χρηματοδότηση και έτσι να δώσουμε και κίνητρα για ε, κατάλληλη κατανομή των συχνοτήτων. Τελευταίο, Νομίζω ότι στην οδηγία θα πρέπει ε, και θα ήταν και χρήσιμο να υπάρχει ένας ορισμός της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και διαδικτυακής ε, ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν σαφείς κανόνες σε θέματα ανταγωνισμού. Η ραδιοτηλεοπτική αγορά είναι μια πολύ ιδιαίτερη αγορά στην οποία κινδυνεύουμε να αλλάξουμε τους δημοκρατικούς μηχανισμούς αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε Ναι. Πιστεύω ότι στο θέμα αυτό, μετά από αυτή την παρέμβαση, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον επόμενο σκιοδησηγητή για την άποψή σας. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως έχουμε συζητήσει επαρκώς και στην συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι συνάδελφοι και στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα επί του οποίου πραγματικά ε, συζητήσαμε και εμβαθύναμε και περνάμε στο εξή. Θα ολοκληρώσουμε με τους κοιόδης και ε, ίσω θα μπορούσε να μιλήσει στη συνέχεια η κυρία Φερχάιεν και η κυρία Καμερέβερτ, διότι μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα τη διαφάνεια, όπω και την κυρία Αντινόλφη, αλλά και όλου. Ο κύριο Ντρογεύσκη έχει ζητήσει το λόγο και μετά ο κύριο Μόργανο και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Φερχάιεν και στην κυρία Καμερέβερτ αν το επιθυμεί. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Έχω μια ερώτηση σχετικά με την εκτίμηση αντικτύπου αυτής της οδηγίας. Οι κανόνες για τις ε, σχέσεις ανάμεσα στους ε, δημόσιους παρόχους και τους ε, ιδιωτικούς είναι κάπως ασαφής. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί μέχρι τώρα που αφορούν τις σύνδρομες κτλ. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν ε, με αφορμή αυτούς τους περιορισμούς θα γίνουν αλλαγές στην οδηγία. Μετά, Νομίζω πως είστε αισιόδοξοι για το ότι θα επιζήσει αυτή η οδηγία και θα είναι σχετική για τα επόμενα 7 χρόνια. Πιστεύω πως ε, θα πρέπει να αρχίσετε ευθύ αμέσω μετά την έγκριση αυτής της οδηγίας να ε, σχεδιάζετε την επόμενη αναθεώρηση. Πιστεύω επίσης πως βρίσκεται πολύ καλές δικαιολογίες για να αποφύγετε να δώσετε λύσεις σε διάφορα δύσκολα θέματα. Τώρα, αυτή η ευελιξία που θα δοθεί στις διαφημίσεις είναι κάτι που δεν με βρίσκει και τόσο σύμφωνο και δεν είμαι αισιόδοξο. Νομίζω πως αυτή η ευελιξία θα χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε οι διαφημίσεις να προβάλλονται την καλύτερη στιγμή για τους παρόχους, για τα κανάλια και όχι για τους ε, θεατές. Επίσης, Ας μην ξεχνάμε ότι οι ραδιοτηλεπτικοί φορείς εκτός Ευρώπης δεν θα έχουν καμία ευθύνη με την παρούσα οδηγία. Ο κύριος Μόρκανο τώρα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σήμερα το πρωί ο γύρος τραπέζης ε, με τις παρεμβάσεις που ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των των συναδέλφων έχουν ε, θέσει τα ε, κύρια θέματα. Εγώ παρεμβαίνω για να πω ότι θεωρώ ότι είναι θετικές οι προτεραιότητες που μας υπέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποιες προσθήκες προφανώς. Ε, από πλευράς μου θα πρέπει να υπολογίσουμε και το ε, συνολικό χρηματικό κόστος, ε, διότι είναι αρκετά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και άρα είναι σημαντικό να γίνει αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μέρημνα όχι μόνο για τις μικρές επιχειρήσεις, ίσως να τις ορίσουμε λίγο καλύτερα, διότι είναι πολλές οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όχι μόνο μικρή ε, κλάδη, αλλά πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα. είναι άλλωστε ένα από τα στοιχεία τα οποία επιτρέπουν ε, ακριβώς ε, να βοηθήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε εμείς στις επιχειρήσεις. Αν δεν υπάρχει κατάλληλη μέρημνα, δεν μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να παραμείνουν στην αγορά. Το άλλο στοιχείο αφορά την ε, δημοσιογραφική ευθύνη για τις πλατφόρμες και νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στο θέμα αυτό, αλλιώς θα υπάρχουν ε, δηλώσεις ε, ε, καλών προθέσεων οι οποίες δεν θα έχουν και καμία συνέχεια. Και υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο το αναφέρω όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων και το θέμα της προσβασιμότητας. Διότι και η προσβασιμότητα είναι θέμα το οποίο μας επιτρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο η πολιτιστική και η δημιουργική βιομηχανία που ενδιαφέρουν σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μόργανο. Ο κύριος Μαλτέζε. Ναι, υπάρχουν αρκετές πτυχές. Πρέπει να πω ότι πέραν των τεχνικών στοιχείων, εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά τη γενικότερη τοποθέτηση. Νομίζω ότι η ανάλυση που γίνεται δεν είναι αρκετά ρεαλιστική για το πώς εξελίσσεται αυτή η αγορά. Φυσικά δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό, γιατί κανένα δεν ξέρει στην πραγματικότητα πώ θα έχουν τα πράγματα σε λίγα χρόνια. Κανεί δεν θα είχε φανταστεί ότι θα είχαμε αυτή την τόσο ταχύ επανάσταση στα μέσα. Πέραν όμως της ευελιξίας που υπενθύμησε η συνάδελφος Φερχάιεν, αλλά και ε, στον τομέα της ενημέρωσης. Οι συνέπειες που είχαν οι τελευταίες τεχνολογικές επαναστάσεις ήταν ε, να ε, καταρρύψει τα πρότυπα ενημέρωσης και μάλιστα με ριζοσπαστικό τρόπο το δίκτυο είναι γεμάτο από πηγές πληροφόρησης, οι οποίες ε, δεν είναι κατάλληλα τεκμηριωμένες και ορισμένες φορές ε, διαχέουν ψευδείς πληροφορίες και μάλιστα αυτό είναι μια μεγάλη επιχείρηση. Υπάρχουν περισσότερες επαφές για ένα μύθο παρά για μια πραγματική ιστορία. Και δεν μπορούμε να βρούμε και ποιος είναι υπεύθυνο. Ε, το ίδιο άρθρο ε, μπορεί να αναρτηθεί στη σελίδα μιας εφημερίδας. Μπορεί να είναι στο facebook στη συνέχεια, μπορεί να αναρτηθεί σε τελείως διαφορετικά ε, στο και αυτό φυσικά έχει τελείως διαφορετική ευθύνη στη συνέχεια. Πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο πιο αποφασιστικοί στον τομέα αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα έπρεπε να αναφέρουμε, όπως για παράδειγμα η διαφήμιση. Επειδή όμω αναφέρθηκε και το θέμα τη κατηγορία για σύγκρουση συμφορώντων για τι δύο συναδέλφου, για την κυρία Φερχάιεν και την κυρία Καμερέβερτ, πρέπει να πω ότι το συζητήσαμε το θέμα αυτό, έγινε και συνέντευξη τύπου, το συζητήσαμε όπως ζήτησα στη συνεδρία των συντονιστών και εγώ προσωπικώς πίστηκα ότι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα σύγκρουση συμφερόντων. Υπάρχει όμως ε, ένα πρόβλημα πολιτικής ε, Ευκαιρία, αν θέλετε, το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο καλύτερα πριν προχωρήσουμε. Διότι μπορεί να επισκιάσει τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε ε, για τη συνέχεια. Και επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, θα έπρεπε ίσως να το συζητήσουμε λίγο ακόμα μέχρι ποιου σημείου είναι θεμητό εάν και δεν συμμετέχει κάποιος σε κάποιο διοικητικό συμβούλιο, αλλά με κάποιο τρόπο εμπλεκόμαστε στη διαχείριση ενός ε, δημοσίου τηλεοπτικού καναλιού, το οποίο υπόκειται και στην ε, νομοθεσία που θα συζητήσουμε. Δηλαδή, αφενός ε, καθορίζονται γενικοί κανόνες και αφετέρου τρόπον την ακόμα και αν είναι με έμεσο τρόπο, χωρί να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων αυτή καθεαυτή, εμπλεκόμαστε στη διαχείριση ενό τηλεοπτικού δικτύου. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι προκειμένου να αποφύγουμε να υπάρχει ένα κλίμα ε, στο οποίο δεν θα υπάρχει επαρκής διαφάνεια, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε λίγο ακόμα και συμφωνώ με την συνάδελφο Αντινόλφη, αν και δεν πιστεύω ειλικρινά ότι οι δύο συνάδελφοι έχουν ε, πραγματικά σύγκρουση συμφερόντων στο θέμα αυτό. Η Πρόεδρος. Να δώσω το λόγο στην κυρία Φερχάιεν και στην κυρία Καμερέβερ, διότι είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση και πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να γίνει δημόσια συζήτηση. Εχθέ όμω ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση λέγοντα ότι δεν θεωρείται ε, ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή και δημόσια η συζήτηση θα μπορέσει να μας ε, βοηθήσει να έχουμε αυτή τη διαφάνεια. Διότι δεν υπάρχει συμμετοχή σε διοικητικό συμβούλιο, σε κάποιο συμβουλευτικό όργανο και εποπτικό όργανο συμμετέχουν οι συνάδελφοι. Επομένως ε, δεν ε, θα ήθελα να συνεχίσω όμως. Θα το δώσω το λόγο στην κυρία Φερχάιεν. ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που συζητήθηκε έντονα χθε. Προσπαθήσαμε και να εξηγήσουμε τι συμβαίνει στην συνέντευξη τύπου την ε, περασμένη Τρίτη. Ε, θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, διότι, αυτό το συμβούλιο, αυτό το το Συμβούλιο δεν είναι εποπτικό συμβούλιο, δεν έχει κανέναν τέτοιο εποπτικό ρόλο, αλλά ε, εκπροσωπεί τους ε, θεατές. Ομαδοποιεί τους ε, θεατές ενός καναλιού, αλλά δεν ε, συμπεριλαμβάνεται κάποιο μέλος κυβέρνησης κτλ. Αλλά είναι ένα σύνολο, μία επιτροπή με που αποτελείται και από ευρωβουλευτέ. Εγώ πιστεύω πως δεν έχει νόημα αυτή, ε, η, αυτό το συμβούλιο. Και λόγω της νομικής βάσης υπάρχει απόλυτη ανεξαρτησία και αυτό το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει ανεξάρτητη χρηματοδότηση. Είναι ανεξάρτητο τελείως από τα κανάλια, από το, από το VDR. Και αυτό αναφέρεται ρητά ότι δεν δίνει αναφορά ούτε στο ΒΕΝΤΕΡ ούτε στην κυβέρνηση της ε, Ρινανίας Βεσφαλίας αλλά η υποχρέωση που έχει αυτό το Συμβούλιο είναι να εκπροσωπεί τους τηλεθεατές και την ίδια υποχρέωση έχουμε και εδώ απέναντι στους ε, θεατές. Πιστεύω λοιπόν πως δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ωστόσο, εάν πολιτικά υπάρχει πρόβλημα το να είναι δύο ε, και οι δύο από τη Γερμανία, τότε θα ήθελα να πω ότι εδώ δεν βρισκόμαστε ως, ε, ως Γερμανοί υπήκοοι, αλλά ως ευρωβουλευτές, οι οποίοι έχουν ε, υπό την ευθύνη τους όχι τους ε, πολίτες μόνο ενός ε, κράτους μέλους, αλλά όλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν ενεργούμε προς το συμφέρον όλων. Και πιστεύω πως η δουλειά μου το έχει δείξει αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Δεν εκπροσωπώ λοιπόν τα συμφέροντα του γερμανικού λαού, αλλά όλες τις, ε, όλων των πολιτών της Ένωσης. Και αυτό σας ζητώ να το λάβετε υπόψη. Εάν λοιπόν ενοχλεί το ότι δύο Γερμανοί πήκοοι είναι συνεισηγητές μιας έκθεσης, τότε Ας μην το κάνουμε αυτό ποτέ ξανά στο μέλλον, να είναι δηλαδή δύο συνεισηγητές από την ίδια ε, χώρα. Σε αυτή την περίπτωση, όμως πιστεύω πως τα πράγματα ε, θα γίνουν πιο δύσκολα και σίγουρα πρέπει να αποφύγουμε να εκπροσωπεί ο καθένα τα συμφέροντα της δικής τους χώρας. Γι' αυτό όμως ε, πιστεύω πως ε, έχουμε και σκιώδεις εισηγητές, υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι συνεισηγητέ και οδησηγητές σε μία έκθεση έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποφία. Αυτό λοιπόν το εξήγησα από την αρχή Ιδιαίτερα σε αυτήν την έκθεση, σε σχέση με τις προηγούμενες, χρειάζεται ακόμα περισσότερη διαφάνεια και διαφάνεια και στις συνομιλίες. Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται και κλεισμένων των θυρών, καμία συνομιλία δεν πρέπει να γίνεται τέτα τέτ, αντίθετα πρέπει να γίνονται ανοιχτές δημόσιες ε, ακροάσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και όλοι να λαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες που λαμβάνουν και οι συμμετέχοντες έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια που πρέπει για να συνεχίσουμε τις ε, διαβουλεύσεις. Αυτές οι συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούλιο και, τον, ε, και τώρα τον Ιούνιο. Μετά τις θερινές διακοπές θα συνεδριάσουμε ξανά, θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων το Σεπτέμβριο, όπου πιστεύω θα είναι αρκετά έντονη αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Είναι μια πολύ καλή προθεσμία. Έχουμε περισσότερο χρόνο από ό,τι για όλες τις υπόλοιπες εκθέσεις. Και ε, θεωρώ ότι τρεις εβδομάδες που έχουμε είναι αρκετός χρόνος έτσι ώστε να μπορέσουμε να κοιτάξουμε ε, με προσοχή το φάκελο και να ε, το να επεξεργαστούμε και να επεξεργαστούμε τις δικές μας προτάσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αλλάξει αυτό το δυσάρεστο κλίμα που έχει δημιουργηθεί με το γεγονός ότι είμαστε συνεισηγήτριες ε, δύο βουλευτές από την ίδια χώρα. Πρέπει να ε, αλλάξει αυτό το κλίμα και εύχομαι με αυτά που μόλις σας είπα να έχει συμβεί αυτό. Ε, πιστεύω πως Θεωρώ, μάλλον ελπίζω, πως έχω κερδίσει την εμπιστοσύνη σας με τη δουλειά που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια και πιστεύω να συνεχίσω να το κάνω. Ευχαριστώ πολύ, Σαμπίνη. Η Πέτρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ. Η Ζαμπίνη Φεχάιεν τα εξήγησε πληρέστατα σχετικά με τις διάφορες μομφές για δίθεν συγκρούσει συμφερόντων. Ούτε και εγώ βλέπω να είναι δεδομένη τέτοια σύγκρουση συμφερόντων, γιατί και ως ευρωβουλευτή αλλά και ως μέλος του ραδιοφωνικού συμβουλίου του σταθμού ARD, που είναι δημόσιο σταθμό στη Γερμανία. Αυτά λέει και ο νόμος για το ARD της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, ότι δηλαδή οι εκπρόσωποι στο ραδιοφωνικό συμβούλιο εκπροσωπούν το δημόσιο συμφέρον των ακροατριών και ακροατών. Όχι τα συμφέροντα του ίδιου του VDR και ότι εμείς έχουμε εκλεγεί για να ελέγχουμε τα όσα πράττει το VDR, η δυτικογερμανική ραδιοφωνία δηλαδή, που έχει δημοσία εντολή και ότι επομένως να εμείς ελέγχουμε ότι εφαρμόζει ορθά την δημόσια εντολή που διαθέτει, χωρίς να έχουμε καμία άμεση επιρροή στο πρόγραμμα του σταθμού. Αυτά είναι ευθύνη της δημοσιογραφικής σύνταξης και του διευθυντού του καναλιού. Σε ό,τι αφορά <clears throat> την πληρωμή, πρόκειται απλώς για επιστροφή δαπανών που προβλέπεται στον ίδιο τον προϋπολογισμό του Ραδιοφωνικού Συμβουλίου. Μάλιστα ψηφίστηκε νέος νόμος που λέει ρητά ότι ο προϋπολογισμός αυτός οφείλει να είναι διαφανής και ανεξάρτητος από τον προϋπολογισμό του ΒΕΝΤΕΡ, του καναλιού δηλαδή ΒΕΝΤΕΡ, που δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωμα συμμετοχής ο ΒΕΝΤΕΡ. Τα χρήματα του προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Συμβουλίου προέρχονται από τα τέλη που πληρώνει ο κάθε ακροατής και κάθε ακροάτρια στην ε, Γερμανία. Έτσι λοιπόν με την έννοια αυτή δεν υπάρχει περιθώριο για σύγκρουση συμφερόντων και αυτά που εξήγησε η Ζαμπίνε Φεχάιεν είναι σωστά. Το Συμβούλιο αποτελείται από 49 άτομα από τα οποία 9 προέρχονται είτε από τοπική Γερμανική Βουλή, Βουλή Κρατηδίου είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως με τη μορφή αυτή και με τη συμμετοχή αυτή δεν έχουμε απολύτως καμία δυνατότητα να κυριαρχήσουμε στην Επιτροπή αυτή του Ραδιοφωνικού Συμβουλίου. Πρόκειται για καθήκον το οποίο μας έχει αναθέσει μάλιστα το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Αυτό αποκλεί οποιαδήποτε κυριαρχία στις αποφάσεις του Ραδιοφωνικού Συμβουλίου. Γνωρίζω ότι έχει ιδιαιτερότητες το σύστημα στη Γερμανία και κατανοώ ότι μπορεί αυτό να οδηγήσει και σε κάποιες παρανοήσεις, διότι γνωρίζω ότι το σύστημα αυτό της δημόσιας ραδιοφωνίας είναι διαφορετικά διαμορφωμένο σε άλλες χώρες μέλη και ότι βεβαίως σε άλλες χώρες μέλη ασκούνται και επιρροές και από τις κυβερνήσεις και από το δημόσιο σε τέτοια συμβούλια. Σας διαβεβαιώ όμως ότι στη Γερμανία υπάρχουν οι νομικές διατάξεις που αποτρέπουν οποιαδήποτε τέτοια δυνατότητα. Και όπου δεν υπάρχουν τέτοιες, έχει φροντίσει με την ομολογία του το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του άλλου σταθμού του ΤΣΕΤΕΦ. Μπορείτε λοιπόν να αισθάνεστε απολύτως ασφαλείς ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ασκηθεί η αδίποτε κυβερνητική επιρροή. Δεν υπαγόμαστε ούτε άλλωστε στο τοπικό κοινοβούλιο, δηλαδή στο κοινοβούλιο της Βόρειας της Βεσσαλίας, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο φορέα. Νομίζω ότι εξήγησα πλήρως την κατάσταση. Η διαδικασία που έχουμε επιλέξει και ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι τίθενται και ερωτήματα και ότι προκαλεί κάποιες επιφυλάξεις το γεγονός ότι δύο Γερμανίδες έχουμε αναλάβει την συνεισήγηση Κάνουμε την προσπάθεια και με τη συλλογική διαδικασία αλλά και με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε επιλέξει να δώσουμε να καταλάβουν όλοι ότι επιθυμούμε απολύτω να συνεργαστούμε με του κοιόδη ηγητέ και συντηρητέ, ότι θέλουμε να είναι απολύτω διαφανής η διαδικασία, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συναντήσουμε ενδιαφερομένου stakeholder στα κρυφά Όλοι οι stakeholder θα πρέπει να γνωρίζουν απολύτως τι έχουν πει οι άλλοι ανταγωνιστές τους ή και συνεταίροι τους. Νομίζω ότι αυτά που λέω είναι λογικά και σωστά. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι στη διάθεσή μας ήδη από την 25η και μπορούμε να δούμε τώρα και μπορείτε να δείτε όλοι τι προτάσεις και ποιες προτάσεις θέλετε να κάνετε. Δεν είναι ανάγκη να καθίσετε να περιμένετε τις σοφίες που θα γράψουμε στο χαρτί εμείς. Ο καθένας μπορεί να αρχίσει να εργάζεται ήδη. Και νομίζω ότι με την 13η δεκάτου που έχουμε βάλει ως προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών, καλά έχουμε κάνει. Θα πω και δύο λέξεις τώρα για το ουσιαστικό περιεχόμενο. Ακερότητα σήματος. Αυτό και εμένα με ενδιαφέρει πολύ, πάρα πολύ μάλιστα, διότι θεωρώ ότι εδώ στην ουσία λείπει, στην πράξη λείπει μια ρύθμιση από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ακερότητα του σήματος, η ακερότητα της εκπομπής πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και να μην μπορεί ο καθένας να παρεμβαίνει και να καταστρέφει το έργο αυτό ή να υποφελείται από πράγματα τα οποία δεν έχει χρηματοδοτήσει ο ίδιος. Το δεύτερο, ο γεωγραφικός αποκλεισμός, το geo-blocking, αυτό δεν είναι θέμα που εντάσσεται στην ε, οδηγία οπτικοακουστικών μέσων, την AVMS, είναι ζήτημα το οποίο μπαίνει στο δίκαιο του δημιουργού και δεν έχει καμιά σχέση εν προκειμένου. Γι' αυτό και εάν θέλουμε να συζητήσουμε το geo-blocking πρέπει να το κάνουμε σε άλλο σημείο, όχι στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας AVMS, που είναι δηλαδή η οδηγία των οπτικοακουστικών μέσων και των σχετικών υπηρεσιών διότι νομίζω ότι εν τέλει, αν γίνει αυτό δηλαδή, θα υπερεπιβαρυνθεί το περιεχόμενο της ε, οδηγίας AVMS. Ευχαριστώ, Μαλτέζε. Θα ήθελα να είμαι λίγο πιο σαφής, γιατί ίσως ε, δεν ήμουν σαφής. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει σύγκρουση ε, συμφερόντων όπως αναφέρθηκε στο άρθρο του Πολίτικο. Και πίστηκα και από τις ε, εξηγήσεις των δύο συναδέλφων, διότι δεν είναι υπάλληλοι της ε, ε, δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και όχι γιατί είναι Γερμανίδες, αλλά διότι συμμετέχουν σε έναν οργανισμό που είναι πολιτικό όργανο στη χώρα τους και με αυτή την έκθεση τους δίνουμε ένα άλλο πολιτικό όργανο, ένα πολιτικό μέσο σε πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ένα πολιτικό ε, πλαίσιο σύγκρουση συμφερέντων. Εγώ δεν γνώριζα τη δομή της γερμανικής τηλεόρασης και ενημερώθηκα για το πώς λειτουργεί. Ας πούμε ότι αυτοί οι οργανισμοί στους οποίους συμμετέχουν οι συνάδελφοι θα μπορούσαν τρόπον τινά να είναι ε, αντίστοιχες με τις εποπτικές επιτροπές που υπάρχουν στην Ιταλία. Έτσι είναι. Εντάξει, ας πούμε ότι έχουν σχέση με τους χρήστες. Εγώ θεωρώ ότι αν εγώ συμμετείχα σε έναν οργανισμό ο οποίος έχει σχέση με την ε, Ιταλική Δημόσια Τηλεόραση, θα ήταν ακατάλληλο να ζητήσω μία έκθεση η οποία ρυθμίζει την ε, Ευρωπαϊκή Δημόσια Τηλεόραση. Και νομίζω ότι είναι ε, ακατάλληλο από πολιτική σκοπιάς. Κατά τα άλλα δεν αμφισβητώ καθόλου την προσωπική εντιμότητα και την οικονομική διαφάνεια των δύο συναδέλφων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ τον κύριο Μαλτέζε, η κυρία Τόμ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω ιδέα πόσο συναισθηματικοί είναι οι συνάδελφοι. Εμείς στην Εστονία προσπαθούμε να ρυθμίσουμε το ζήτημα και προσπαθούμε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά όταν λέμε ότι πρέπει να επιλέξουμε ποιοι θα πρέπει να εκπροσωπούν τους χρήστες, τους θεατές ε, θα πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη ισορροπία και σε γεωγραφικό επίπεδο και σε άλλα επίπεδα. Επομένως θα ήθελα να κάνω μια πρόταση για το μέλλον ώστε να το ρυθμίσουμε αυτό με ήρεμο τρόπο. Ας συνεχίσουμε με την έκθεση αυτή, όπως ε, ε, μέχρι τώρα. Κανείς δεν είπε ότι υπάρχει κάποια παραβίαση. Ίσως θα μπορούσε να υπάρχει βιοντολογικό θέμα, αλλά πιστεύω ότι αν ε, ε, πούμε την άποψή μας, μπορούμε να ρυθμίσουμε και το δεντολογικό ζήτημα. Η πρότασή μου είναι να φροντίσουμε να υπάρχει γεωγραφική ισορροπία, όχι μόνο για τις ακροάσεις, αλλά όταν έχουμε και συνεισηγητές. Και πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε τέτοιο πρόβλημα εάν οι συνάδελφοι ευθύ εξ αρχής είχαν δηλώσει ότι έχουν και αυτά τα καθήκοντα ε, στους οργανισμούς αυτούς. Η κυρία Τρούπολη. Ναι. Επειδή εγώ ανήκω σε μια μικρή πολιτική ομάδα, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιε από τι ε, μικρότερε πολιτικέ ομάδε ε, δυσανασχετούν για την κατάσταση. Θα ήθελα να επενθυμίσω όχι τη χθεσινή συνεδρία των συντονιστών, αλλά την προηγούμενη συνεδρία των συντονιστών, όταν συζητήθηκε το θέμα και ήταν σαφέ ότι οι δύο μεγάλε πολιτικέ ομάδε εξακολουθούν να έχουν του περισσότερου βαθμού, ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό και ξέραμε ότι υπάρχουν άτομα τα οποία είναι και γνωσμένου κύρου ε, επί των θεμάτων αυτών. Εγώ προέδρευα τότε στην ε, συνεδρίαση και ήταν απόλυτα σαφές ότι ακόμα και αν υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι ε, υπάρχει μια δυσαρέσκεια για την κατάσταση, υπήρχε μια πλειοψηφία στην ψηφοφορία που έδωσε την ε, έκθεση στις δύο αυτές μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες γιατί υπάρχει το σύστημα της βαθμολογίας. Εφαρμόστηκε το σύστημα αντεχών που εφαρμόζεται πάντα όσον αφορά την ε, πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι προφανώς υπάρχει διαφορετική νομοθεσία στα κράτη-μέλη όσον αφορά τις δημόσιες ε, τηλεοράσεις. Στη Γερμανία, και αυτή είναι και μια πρόσφατη αλλαγή, είναι σαφές ότι αυτός ο οργανισμός είναι ένας ειδικό οργανισμός, ένας ανεξάρτητος εποπτικός οργανισμός, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με Δικοτικό Συμβούλιο Επιχείρησης. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση, διότι Ιδάλω, πράγματι θα υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Αν ήταν ένα διοικητικό συμβούλιο, το είπα χθε για παράδειγμα, το ε, ε διοικητικό συμβούλιο τη Volkswagen ή τη Mercedes ή οποιοδήποτε άλλο. Αλλά δεν έχει σημασία. αυτό ο εποπτικό οργανισμό στόχο έχει να ελέγχει τη δημόσια αποστολή του δικτύου. Εάν δηλαδή εφαρμόζουν την αποστολή του προγράμματος όπως θα έπρεπε και αν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφόρον. Οι πολιτικοί που συμμετέχουν σε αυτό τον ανεξάρτητο υποπτικό φορεία δεν έχουν την πλειοψηφία. Οι άλλε ομάδε, η ομάδα τη κοινωνία των πολιτών είναι αυτέ οι οποίε πλειοψηφούν και επομένω δεν θα πρέπει να γίνεται σύγκριση με διοικητικά συμβούλια. Η εντύπωση μου λοιπόν ήταν ότι επειδή ήταν σαφές ότι υπάρχουν κάποιες εντάσεις στην Επιτροπή μας, ο καλύτερος τρόπος να το λύσουμε είναι να εργαστούμε με όσο το δυνατόν πιο διάφανο τρόπο. Αυτό το έχουμε ήδη ανακοινώσει. Επομένως θα προσπαθήσουμε να γίνονται κοινέ συνεδριάσεις, να μην γίνονται διαζώσεις συνεδριάσεις για να μπορούμε να αποφασίσουμε. Και εκεί θα δείτε ότι υπάρχει μια διάθεση εμπιστοσύνη και καλή ε, συνεργασία, διότι εγώ όταν προσωπικώς ε, το ήλεγξα δεν διαπίστωσα ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ίσως για το μέλλον λοιπόν θα ήταν καλύτερο να δούμε εάν μπορούμε να έχουμε μια άλλη μορφή ισορροπία. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει ε, να βασιστούμε στην υπόσχεση ότι θα είμαστε απόλυτα διάφανοι και θα συνεργαστούμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ για την σαφήνεια και για αυτή την ανταλλαγή απόψεων, διότι τελικά έγινε επανάληψη της χθεσινής συζήτησης, αλλά δικαίως έγινε αυτή η επανάληψη και καλό είναι που γίνεται και δημοσίως και με διαφάνεια. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που είπε η Αντιπρόεδρος κυρία Τρούπελ. Την ευχαριστώ και για τη διευκρίνηση, ευχαριστώ και τις συναδέλφους και αντιλαμβάνομαι απόλυτα και το αίτημα του κυρίου Μαλτέζε που ήταν διτό. Το ένα αναφερόταν στη σύγκρουση συμφερόντων, για το οποίο και εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι δεν τίθεται, γιατί αλλιώ δεν θα είχα προχωρήσει προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία βάση, για δύο λόγου. Καταρχά, ότι δεν υπάρχει ε, καμία συμμετοχή σε οργανισμό διαχείριση. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη αρχή, την οποία ορίζει το Κοινοβούλιο, αποτελείται από 50 μέλη. Ένα μικρό ποσοστό είναι εθνικοί και ευρωπαίοι βουλευτές και γιατί και η αποζημίωση των εξόδων γίνεται επί τη βάση ενό ανεξάρτητου προπολογισμού και όχι από τον προπολογισμό τη τηλεόραση. και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ε, δούμε κατά πόσον μπορεί να στοιχειοθετείται πράγματι σύγκρουση συμφερόντων. Επίση, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, όπω γίνεται πάντα, η επίσημη απόφαση για το ποιες ήταν οι πολιτικές ομάδες ε, στις οποίες θα πρέπει να ανατεθεί η έκθεση και Έχουμε και τους ε, συνεισηγητές οι οποίοι επικυρώθηκαν από το Προεδρείο ε, την Πέμπτη και αποφασίστηκε ότι θα έχουμε εισηγητές από τις δύο πολιτικές ομάδες, από το ΕΛΚ και τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Να υπενθυμίσω ότι οι δύο συνάδελφοι όχι μόνο είναι εμπειρογνώμονες, αλλά είναι και συντονίστριες των πολιτικών της Επομένως, ε, είναι πολύ σημαντικό και αυτό εντός των πολιτικών ομάδων και αποφάσισαν οι πολιτικές ομάδες. Και αυτές οι αποφάσεις, όπως ξέρετε, γίνονται... Διακόπτε, κύριο Μαλτέζε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση. Κανείς δεν αμφισβητεί την επιλογή. Εμείς δεν επιλέξαμε τα ονόματα, επιλέξαμε τις πολιτικές ομάδες. Δεν λέει κανείς ότι το και οι σοσιαλιστές και οι δικομάτια. Ναι, επιτρέψτε μου, λέει ο Πρόεδρος, να σας κάνω απλώς έναν απολογισμό της κατάστασης για να δείτε τι έγινε. Συλλογικά και οι ομάδες εκφράζουν την άποψή τους, γιατί οι πολιτικές ομάδες υπέδειξαν τι συναδέλφουν ως εισηγήτριες. Θεωρώ ότι αυτό που έθεσε η κυρία Τινάλφη και ο κύριος Μαλτέζε ίσως λίγο πιο αναλυτικά. Πρέπει να το προσέξουμε υπό την έννοια ότι και εγώ πάντα, αγαπητοί συνάδελφοι Τόμ, ε, θεωρώ ότι αν μπορούμε να έχουμε καλύτερη γεωγραφική κατανομή, ε, καλό είναι να το κάνουμε. Αλλά αυτή τη φορά επέλεξαν οι πολιτικές ομάδες ελεύθερα και για τη σημασία αλλά και για την αξία των συναδέλφων. Και αυτή τη στιγμή λέμε και εμείς ότι ο καλύτερος τρόπος να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανοιχτοί και από γεωγραφική και από πολιτική σκοπιά και από πλευράς διαφάνειας και ενώπιον των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη μέθοδος εργασίας, να γίνονται δημοσίως τα πράγματα, υπάρχουν τρεις συνεδριάσεις οι οποίες προβλέπονται με τους διάφορους ενδιαφερομένους και φυσικά και η πολιτική και προσωπική ε, δεοντολογία των συναδέλφων και εδώ σα διαβεβαιώ και εγώ ότι θα γίνει σεβαστό από πλευρά μου ως πρόεδρος και φυσικά να συνειδητοποιήσουμε όλοι όπως είπαν και η Πέτρα και η Σαμπίνε, ότι όλοι δεσμευόμαστε να είμαστε ε, επάξιοι εκπρόσωποι των πολιτών. Δεν είμαστε μόνο αιρετοί, αλλά είμαστε εκπρόσωποι των πολιτών μας. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι επιβεβαιώνεται η ε, ανάθεση της έκθεσης εσάς και ε, να συνεχίσουμε τώρα τη συζήτηση και για λόγους ευγενίας προς τις ε, προσκεκλημένες μας. Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά πρέπει να είναι απόλυτα σαφές το ζήτημα σε όλα τα θεσμικά επίπεδα. Δεν ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Ε, α, ο κύριος Γραμματικάκης, παρακαλώ. Εγώ νομίζω κυρία Πρόεδρος ότι είναι πολύ σωστά αυτά που είπατε και δεν θα έπαιρνα το λόγο αν δεν έβρισκα ένα άλλο κίνδυνο. Να ζήσουμε το λέω και για τη Σαμπίνα και για την Πέτρα, την απόλυτη ηθική τους, ε, θα έλεγα, καταξίωση. Αλλά ο κίνδυνος είναι να ζούμε συνεχώς υπό το φόβο κάποιας κατηγορίας που εκτοξεύεται δεν ξέρω από πού. Τα κοινωνικά δίκτυα οργιάζουν στις συκοφαντίες και κατά κάποιο τρόπο θα ερχόμαστε εδώ στις συνεδριάσεις αποστηρωμένοι, χωρίς επαφή με την πραγματική ζωή. Αυτός είναι μεγάλος κίνδυνος γιατί μην ξεχνά κανένας ότι οποιαδήποτε γνωμοδότηση, οποιαδήποτε εδώ συζήτηση, εάν υποτεθεί ότι κάποια συμφέροντα δεν τα καταλαβαίνω αυτά και πολλοί, ανοησίες είναι, ε, προσπαθούν να επικρατήσουν, φύγει και εμάς τους ίδιους που κάνουμε προτάσεις, που είμαστε στιώδεις και μη στιώδεις. Θα πω λοιπόν να σταματήσει αυτή εδώ η συζήτηση. Ε, Φοβάμαι πάρα πολύ παρόμοιες συζητήσεις. Είμαι απολύτως, ε, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις δύο συναδέλφους, στην Πέτρα και στην ε, Σαμπίνα και ξέρουν πολύ καλά οι δύο και οι πέντε και οι δέκα ότι όταν χρειαστεί να κάνω τολμηρές παρατηρήσεις δεν φοβάμαι κανένα. Εγώ κυρία Πρόεδρος το δηλώνω, είμαι αντιπρόεδρος στη δημόσια λυρική σκηνή της Ελλάδος. Και αν μια στιγμή ψηφίσετε ότι ο Βάγνερ είναι ο καλύτερος συνθέτης φοβάμαι ότι θα κατηγορηθώ εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή σήμερα είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής ε, προς τιμήν του Βάγνερ ε, αλλά και όλων των υπολείπων, ε, το Βέρντι μην ξεχάσουμε, το Σούμαν κλπ. Γιατί αλλιώ ε, ε, ελοχεύει ο κήτος να θεωρήσουν ότι υπερασπιζόμαστε μόνο τη χώρα μα. Θα ήθελα λοιπόν με αυτή την ευχάριστη νότα να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, αλλά φυσικά αυτό πρέπει να το φροντίσει και όποιος κάνει δηλώσεις στο, στον τύπο οι οποίες ε, δεν έχουν βάση. επειδή εγώ σε μια προηγούμενη ζωή μου ήμουν δημοσιογράφος, ε, ξέρω ότι πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη δημοσιογραφική δεοντολογία. Να ε, ολοκληρώσουμε λοιπόν με το θέμα αυτό για να συζητήσουμε αυτή την οδηγία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελευθερία και αμοιβαίο σεβασμό σε κλίμα συνεργασίας. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα μόνο, διότι θα ήθελα να ε, ε, μου διευκρινίσετε κάποια σημεία. Νομίζω ότι όλοι οι συγητές, και όλοι οι συγητές, οι συνάδελφοι εξέφρασαν την άποψή τους, ε, κάλυψαν όλα τα θέματα και θα ήθελα να μου πείτε για το θέμα της διαφάνειας, ε, της διαφήμισης συγγνώμη, και της ευελιξίας που ζητούμε. Αυτό φυσικά προκύπτει από την ανάγκη ισορροπίας ε, των πόρων. Και το είπαν και οι συνεχέτριες, ε, θα έπρεπε ίσως να εμβαθύνουμε και λίγο στο γεγονός ότι Αυτές οι πλατφόρμες ε, του video on demand ε, και των υπηρεσιών on demand θα πρέπει να συμμετέχουν λίγο περισσότερο και να ε, μην είναι τόσο παρασιτικός ο ρόλος τους όπως είναι σήμερα, διότι ξέρουμε ότι αυτά στην πραγματικότητα δεν διατίθενται δωρεάν, είναι πώληση για διαφήμιση των προφίλ των χρηστών. Θα πρέπει λοιπόν είτε άμεσα είτε έμεσα να συνεισφέρουν στην παραγωγή ευρωπαϊκών έργων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τη διαφήμιση και αυτή την περιβόητη ευελιξία, θα ήθελα να ξέρω τι προκύπτει από τις παρεκκλήσεις για το θέμα αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν ε, κάποιες εξαιρέσεις στο κείμενο ναι, ναι. κάποιων περιπτώσεων. Παραδείγματος χάρη εκπομπές που έχουν ε, πολλούς ανηλίκους θεατές. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Όντως υπάρχει αυτορύθμιση υπό την έννοια ότι ε, αλλιώς χάνονται θεατές. Αλλά το άλλο θέμα αφορά τη σύγχυση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της διαφήμισης, η οποία δεν θα πρέπει να έχει σχέση με το περιεχόμενο, ε, σε σχέση με την προώθηση, τη χορηγία και όλα αυτά τα οποία ε, εντάσσονται στην εκπομπή και ε, ας πούμε ότι είναι και κρυφή διαφήμιση ή είναι ε, ένθετη στο περιεχόμενο. Θα ήθελα λοιπόν να είναι ανοιχτό τελείως το θέμα ή αν υπάρχουν κάποιοι πιο αυστηροί κανόνες από αυτού, διότι αλλιώς οι εκπομπές μετατρέπονται σε τεράστια διαφημιστικά σποτ. Και η άλλη ερώτηση αφορά το θέμα του περιεχομένου που παράγεται από πλατφόρμες ε, ε, όπως το YouTube ή άλλες πλατφόρμες ε, που προωθούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές. Ε, νομίζω ότι στα θέματα αυτά έχουμε επεκτείνει τα θέματα προστασίας για τους ανηλίκους και τη ρητορική μίσους, αλλά θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο ευαίσθητοι σε θέματα όταν υπάρχουν ε, οργανώσεις που ε, παράγουν περιεχόμενο και θα πρέπει να δούμε λίγο περισσότερα πράγματα όσον αφορά την ευθύνη και να μην υπάρχει ευθύνη μόνο για το ε, για το e-commerce ε, και να καλύπτουμε μόνο του ανηλίκου. Να σα δώσω το λόγο γιατί μα πιέζει και ο χρόνο για να απαντήσετε. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και όλου εσά για τι παρεμβάσει σα. Πολλέ ερωτήσεις έγιναν. Δεν θα καταφέρω πιστεύω να απαντήσω σε όλες, όμως θα σταθώ σε τρει-τέσσερι που έχουν άμεση σχέση με αυτό που ε, έχω να πω. Καταρχάς, ερωτήθηκε από πολλούς για τη σχέση ανάμεσα σε γραμμικές και μη γραμμικές εκπομπές και ότι είναι θολά τα όρια. Ε, όπως είπατε και εσείς, εξελίσσονται ταχύτατα τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το στάδιο είναι πολύ δύσκολο να γίνει πλήρης γράμμιση. Όπως είπα και στην αρχή, τα πράγματα αλλάζουν, εξελίσσονται και τα επιχειρηματικά μοντέλα διαφέρουν. Ε, σε αυτές τις δύο ε, περιπτώσεις. Το θέμα είναι πώς θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο μας δεδομένων αυτών των διαφορών στα επιχειρηματικά μοντέλα. Πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές οι στόχοι είναι παρόμοιοι, όμως το θέμα είναι πώς θα προσαρμόσουμε, με την, ε, πώς θα προσαρμόσουμε την νομοθεσία και τι θα κάνουμε. Διαφήμιση γιατί δεν έχει επεκταθεί ε, στην ε, διαφήμιση στις ε, διαδικτυακές πλατφόρμες η νομοθεσία. Το θέμα είναι να δούμε τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, για παράδειγμα θέμητες εμπορικές πρακτικές. Ας δούμε την αντίστοιχη οδηγία με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά, νομίζω πως υπάρχει αρκετά μεγάλο ποσοστό αυτορύθμισης και έχουν δείξει οι ερευνές μας ότι έχει θετικά αποτελέσματα. Αυτή λοιπόν ήταν η αφετηρία μας και γι' αυτό δεν προτείναμε συγκεκριμένη νομοθεσία γι' αυτό. Τώρα σχετικά με τις ποσοστώσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι για την περίπτωση του video on demand υπάρχουν δύο ε, πτυχές. Υπάρχει και το 20% αλλά και η προβολή των ευρωπαϊκών έργων. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ορατότητα αυτών των ευρωπαϊκών έργων στις ε, πλατφόρμες Video On Demand. Τώρα, ε, κυρία Πρόεδρε, με ρωτήσατε για τις πλατφόρμες ε, Video Sharing. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ακριβώς διότι οι χρήστες είναι εκείνοι που κατά μεγάλο ποσοστό δημιουργούν το περιεχόμενο που ανεβάζουν. Υπάρχουν λοιπόν ευθύνες των χρηστών για το τι ανεβαίνει εκεί. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβάλλουμε σχετικέ ποσοστώσεις. Αυτό φυσικά μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά αυτή είναι η διαφορά. Κάτι που ήθελα να τονίσω και έχει σχέση με αυτό που είπατε, είναι ότι επιμένουμε για πλήρη διαφάνεια. Συνεχίζουμε να επιμένουμε. Νομίζω η κυρία Τρούπελ το είπε αυτό στην παρέμβασή της για την έμεση τοποθέτηση και προώθηση προϊόντων, το product placement είναι σαφές ότι εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση πρέπει να ε, αναγράφεται. Αυτά περί διαφάνειας και γι' αυτό λοιπόν μέσω των διτάξεων για τη διαφάνεια ελπίζω να καταφέρουμε να το ρυθμίσουμε. Τώρα, αρκετοί αναφέρθηκαν στην σχέση με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Νομίζω πως εδώ προσπαθήσαμε να καταφέρουμε ένα ελάχιστο ποσοστό ευθύνη για τις πλατφόρμες video sharing. Επαναλαμβάνω, είναι διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο αυτό του video sharing και δεν νομίζω πως χρειάζεται να αλλάξει ε, το καθεστώς ε, ευθύνης. Πρέπει να ε, αυξηθεί η ευθύνη, να, υπάρχει, να υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις και εάν αυτές δεν τηρούνται να υπάρχουν κυρώσεις. Δεν νομίζω όμως ότι πρέπει να αλλάξει το περιεχόμενο, διότι οι χρήστες είναι εκείνοι που κατά μεγάλο ποσοστό το δημιουργούν. Τώρα, πολλοί ε, χρήστες ε, όταν δεν είναι ικανοποιημένοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα κάποιας προσφυγής. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην ε, μεγαλύτερη ευθύνη αλλά μέχρι ένα, που, να, να μην ξεπερνά το όριο. Τώρα, ε, αναφερθήκατε στην, στην προσβασιμότητα και στο Accessibility Act. Πιστεύω πως εδώ ξεφεύγουμε και πάμε πολύ ε, πιο πέρα από τις διατάξεις του άρθρου 7 της, ε, του κανονισμού για την προσβασιμότητα. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν καλύψει η νομοθεσία για την προσβασιμότητα το θέμα αυτό, πρέπει να το κάνουμε εδώ, στην οδηγία. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εμείς θέλαμε να είμαστε συνεκτικοί, να υπάρχει μία συνέχεια και δεν θέλαμε να αλλάξουν ή να επιβραδυνθούν οι διαπραγματεύσεις. Τέλος, για το, την ακαιρεότητα του σήματος και για την δυνατότητα ανείχνευσης. Θα σας παραπέμψω στην αιτιολογική σκέψη 38 που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αναλάβουν ε, εθνική δράση. Εδώ τσακωθήκαμε με την νομική υπηρεσία για να το καταφέρουμε, όμως κατανοήσαμε το πόσο σημαντικό πολιτικά είναι αυτό για την Επιτροπή αυτή. Υπάρχει μια υποχρέωση η οποία θα καλύπτει και, τους, ε, και άλλους ε, παρόχους ε, περιεχομένου. Ξεφεύγει δηλαδή από το πεδίο εφαρμογή. Κάναμε λοιπόν ό,τι μπορούσαμε δεδομένων των νομικών περιορισμών που είχαμε. Όσον αφορά τώρα την ακαιρεότητα σήματος, η κυρία Κάμερ Εύερτ, αν δεν κάνω λάθος, είπε ε, πως αναρωτιέται αν είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ακαιρεότητας σήματος. Επαναλαμβάνω, κατανοώ τις ανησυχίες σας, όμως δεν ξέρω αν αυτή εδώ η οδηγία είναι ο κατάλληλος χώρος για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε το κλείσω θα ήθελα να επαναλάβω ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, προχωρήσουμε γρήγορα. Πιστεύω όχι μόνο για εμάς αλλά και για εσάς. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παροτρύνω να προχωρήσετε σε μια επί της ουσίας συζήτηση έτσι ώστε να, μπορούμε, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ και στην κυρία Πιούρ και στην κυρία Λόνσο για αυτή την πρώτη συνάντηση. Όπως ε, σας είπα, δεν θα είναι η πρώτη, θα είναι η πρώτη από πολλές συνεδριάσεις που θα κάνουμε και η Επιτροπή μας ε, θα είναι ιδιαίτερα δραστήρια. Θέλουμε πραγματικά να εμβαθύνουμε στα θέματα αυτά. Πρόκειται για θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, στρατηγική σημασία και από πλευρά μα η οδηγία αυτή είναι μία από τους πυλώνες της νέας ε, ψηφιακής στρατηγικής, διότι άπτεται του ε, πολιτιστικού περιεχομένου, της ε, πολυφωνίας, ε, αλλά και της προσοχής στις ευρωπαϊκές παραγωγές και στην κυκλοφορία των έργων με ισορροπημένο τρόπο και όπου μπορούμε χωρίς διάκριση μεταξύ γραμμικής και μη γραμμικής υπηρεσίας και να επεκτείνουμε αυτές τις υποχρεώσεις οι οποίες δεν γίνονται σήμερα σεβαστές στα πλαίσια της διαδικτυακής επικοινωνίας και για τους ανηλίκους αλλά και για την ε, ρητορική μίσους και όλες τις μορφές ε, ε, περιεχομένου που δεν είναι αποδεκτό αυτή τη στιγμή. Πρέπει να εργαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Το Κοινοβούλιο φυσικά έχει ένα χρονοδιάγραμμα αρκετά ε, σαφώς καθορισμένο και πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι, οι σκιώδεις συγητές και οι συγητέ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν ώστε το κείμενο το οποίο θα έχουμε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα σε ε, κάποια από τα θέματα τα οποία προέκυψαν και από τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σα. Ζητούμε συγγνώμη αν ε, άλλαξε λίγο και το θέμα τη συζήτηση. Έτσι γίνεται όμω με τις δημόσιες ε, συζητήσει. Ήταν σημαντικό το θέμα και μα βοήθησε να διευκρινίσουμε λίγο καλύτερα και τη θέση τη Επιτροπή μα. Σα ευχαριστώ be in touch. Bene, ora inviterei subito perché siamo in leggero ritardo. Τώρα, επειδή έχουμε καθυστερήσει λίγο, θα ήθελα να καλέσω μια πολύ αγαπητή προσκεκλημένη μας. Allora, prego, accomodatevi. Περάστε, καθίστε. Eh, Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά Έχουμε λοιπόν εδώ μαζί μα. παρακαλώ του συναδέλφου ε, να καθίσουν και να παραμείνουν διότι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και πρέπει να το προσέξετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ. Καθίστε παρακαλώ. Γραμματικάκη. Κυρία Γραμματικάκη, κυρία Φερχάιεν. παρακαλώ. I would like that some colleagues uh, uh, stay here because it's very... Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να παραμείνουν γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον ε, το θέμα αυτό για να συζητήσουμε για τη σύμβαση της ε, UNESCO για την ε, προστασία και την πρόθεση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων. Έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ μαζί μας και πραγματικά μας ενδιαφέρει να γίνει αυτή η συνάντηση τους εκπροσώπους της ε, UNESCO, τον Φραντσέσκο Μπανταρίν και την Τανιέλ Κλής ε, που είναι εδώ και τους ευχαριστούμε. Αποτελεί πολύ σημαντική ευκαιρία για μας. Ε, βέβαια κλείνει ένα πρωινό αρκετά έντονο, είχαμε ψηφοφορίε παρεμβάσεις, συζητήσεις πολύ σημαντικέ, αλλά πραγματικά θέλαμε να μην ε, χαθεί αυτή η ευκαιρία και σα ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας εδώ. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η UNESCO, διότι αυτή τη διετία συναντηθήκαμε αρκετές φορές με την UNESCO και στην Επιτροπή μας, ιδίως ε, η Γενική Γραμματέα, την κυρία Μπόκοβα και ε, τώρα έχουμε τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και έχουμε και τη δυνατότητα να συζητήσουμε ε, μία από τις πιο σημαντικότερες συμβάσεις της UNESCO, του, η σύμβαση του 2005, έχει κυρωθεί από 140 χώρες πλέον, αλλά την έχει κυρώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ε, και χαίρομαστε γιατί ε, υπάρχει νομική βάση στη συνθήκη και μπορούμε να κυρώνουμε συμβάσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις συμβάσεις είναι περισσότερο δεσμευτικές για μας. Ε, η σύμβαση αυτή είναι μια σύμβαση η οποία για πρώτη φορά προβλέπει μια πραγματική σχέση για την ε, συνολική εφαρμογή των θεμάτων αυτών και χαιρόμαστε που είστε εδώ διότι ε, τρόπον τεινά αυτό επικυρώνει την ε, ε, δέσμευση των κρατών μελών και μπορούμε να επαληθεύσουμε κατά πόσον υλοποιούνται αυτοί οι στόχοι που έχετε εντοπίσει. Τι εφαρμόζεται ε, από πλευρά σύμβαση και από πλευρά χωρών μελών αλλά και από πλευρά Ευρώπη. Υπάρχουν αυτοί οι τέσσερι στόχοι υποστήριξη των ε, συστημάτων ε, της ε, διακυβέρνησης για τον πολιτισμό. Και μάλιστα εδώ επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και μια κρίση πόρων, αρχίζουν κάποιες χώρες σιγά σιγά να ξανασκέφτονται το ζήτημα, κυρίως η χώρα μου που αρχίζει να επενδύει πλέον στον πολιτισμό και η Επιτροπή μας είχε και μία πολύ σημαντική έκθεση, την έκθεση Διακόμο για την ε, ολοκληρωμένη διακυβέρνηση και μία ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διακυβέρνηση της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θέμα της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των πολιτισμικών περιεχομένων, η συνεισφορά του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη και το πολύ σημαντικό στόχο της ελευθερίας και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και τα πολιτισμικά δικαιώματα είναι αναπόσπαστο τμήμα των θεμελιωδών των και για πρόσβαση στον πολιτισμό και για την ενεργό συμμετοχή και τη γνώση τη πολιτιστική μα κληρονομιά. Δεν θα επεκταθώ γιατί μα πιέζει ο χρόνο. Απλώ να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλουμε να έχουμε συναχή επαφή μαζί σα. Το Κοινοβούλιο υλοποίησε και ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την UNESCO και χρηματοδότησε ε, εντός του 2016 και ζητάμε και χρηματοδότηση και για το 2017 ένα έργο για τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τους δεσμούς, να υπάρχει ένα δίκτυο και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ε, ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και UNESCO και ε, υπάρχει δέσμευση από το Κοινοβούλιο μας για το θέμα της καταστροφής επίφυσης της πολιτισμικής κληρονομιάς και θα ήθελα να ζητήσω από τις σχόλες να ε, δραστηριοποιηθούν γιατί ε, μόνο εμείς έχουμε στείλει την task force ε, στην αρμόδια υπηρεσία της UNESCO και θέλουμε να έχουμε προστασία των πολιτιστικών αγαθών που η Ευρώπη προσπαθεί να διαφυλάξει βάση και τη σύμβαση. Να σας δώσω αμέσω το λόγο γιατί έχουμε μόνο μισή ώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που καλέσατε μένα και τον συναδελφό μου, κύριο Κλής, εδώ. Για να σας παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή. Όπως είπατε και εσείς, είναι μέρος ε, μιας συνεχιζόμενης δράσης. Η UNESCO και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια ανέπτυξαν ένα πολύ ε, στενό δίκτυο ανταλλαγή ε, πληροφοριών και συνεργασίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που μας καλέσατε. Η μελέτη λοιπόν, η έκθεση που θα σας παρουσιάσουμε, ε, έχετε λάβει νομίζω και εσείς αντίτυπο. Και να σας πω ότι μπορείτε να βρείτε την έκθεση και στο διαδίκτυο. Μπορείτε να βρείτε και μία περίληψη που νομίζω πως θα χρησιμεύσει πάρα πολύ στα μέλη της Επιτροπής. Επίσης, να σας πω ότι μας βοήθησε και η κυβέρνηση της Σουηδίας και το ειδικό τμήμα που ασχολείται με την πολυμορφία. Τώρα, θα ήθελα να πω ότι η έκθεση αυτή ασχολείται με έναν τομέα συνεργασίας ιδιαίτερης σημασίας. Έχουμε κοινού στόχους. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ε, έκφραση της πολυμορφίας μέσω του πολιτισμού. Η πολιτισμική διάσταση, μάλιστα, είναι κάτι που έχει που είναι καθολικά αποδεκτό. Ας μιλήσουμε λοιπόν για κάποιες ε, ιδιαίτερες λεπτομέρειες που μας επιτρέπουν να εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές σε μεγαλύτερη κλίμακα. Τώρα, από την αρχή το project αυτό στηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε μία ε, ομάδα που ασχολήθηκε με την εφαρμογή από το 2010 μέχρι το 2015 είχαμε προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο δολάρια έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις σε 13 χώρες μέσω της κατάρτισης να μπορούν να διαχειρίζονται τις, τις αγορές πολιτισμικών αγαθών και να κατανοήσουν το πώς ε, αλλάζουν έτσι ώστε να μπορούν να χαράξουν αντίστοιχα την ε, πολιτική τους. Τα αποτελέσματα είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μας. Θέλουμε να συνεχίσει η συνεργασία μας, αλλά ε, να σας πω πως ε, παρά το γεγονός ότι έχουμε δικούς μας πόρους, φυσικά δεν θα λέγαμε όχι σε ε, πρόσθετους, και, πρόσθετους πόρους και δεν θα λέγαμε επίσης όχι και στη στήριξη από όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς. Και χάρη στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελπίζω να έχουμε καλά αποτελέσματα. Μέχρι τώρα έχουν προσχωρήσει στη Σύμφωση 144 κράτη-μέλη και χάρη στις προσπάθειες της Ένωσης ε, καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτούς τους αριθμούς. Δεν έχουμε, βέβαια ακόμα, δεν έχουμε βέβαια ακόμα καθολική αποδοχή, όμως ελπίζουμε να φτάσουμε προς εκεί. Τώρα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και δεν θα αναφερθώ στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, όμως βλέπουμε ότι πάρα πολλέ χώρε τώρα έχουν συγκεκριμένη πολιτική για πολιτισμική δραστηριότητα και τα πολιτισμικά αγαθά εξαιτία αυτής της δράσης που στηρίξατε και εσεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, πρώτη φορά σε 10 χρόνια κάνουμε μια τέτοια παρουσίαση εδώ. Τα τελευταία δέκα χρόνια, από τότε δηλαδή που εγκρίθηκε η σύμβαση μέχρι τώρα, έχει αλλάξει δραματικά το πολιτισμικό τοπίο στον κόσμο. Τώρα υπάρχουν ε, εταιρείε ε, κολοσσή στο διαδίκτυο, υπάρχει το ψηφιακό περιεχόμενο, αλλάζει δηλαδή ριζικά ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται, διανέμεται και καταναλώνεται το ψηφιακό πολιτισμικό περιεχόμενο. Κάτι που συζητήσατε και πιο πριν. Εμείς θέλουμε να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον νέο κόσμο. Η έκθεση μας λοιπόν εξετάζει τις εξελίξεις των τελευταίων δέκα ετών, εντοπίζει τα αδύναμα σημεία και τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα του συστήματος. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές καινοτόμε δηλαδή πολιτικές οι οποίες ε, μπορούν να διαχειριστούν και να χειριστούν αυτή την επανάσταση. Κάτι που δεν είναι εύκολο φυσικά, όπως γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, διότι είναι πολύ δύσκολο να μετρήσουμε και τις επιπτώσεις με ποσοτικό τρόπο. Επίσης, θέλουμε αυτές οι πολιτικές να ε, συμπεριληφθούν στην ε, ατζέντα των Ηνωμένων Αθηνών για το 2020-2030. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να συμπεριληφθούν θέματα πολιτισμού, πολιτισμικής κληρονομιάς κτλ. Ε, στην ε, ατζέντα αυτή. Μέχρι τώρα έχει γίνει καλή δουλειά. Τα αποτελέσματα όμως θα τα δούμε και αργότερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείτε μέχρι να τελειώσει το 2016 το αστικό θεματολόγιο το οποίο έχει λάβει υπόψη του πολλά από, πολλές από τις ε, συστάσεις μας. Τώρα, η σύμβαση αυτή έχει ένα ευρύτατο φάσμα στόχων και είναι εύλογο να προκύψουν και ερωτήματα. Πώς δηλαδή η σύμβαση αυτή θα εμπνεύσει οι διάφορες χώρες να αλλάξουν την πολιτική τους, πώς θα εφαρμόσουν την πολιτική αυτή που θα ε, αλλάξει, πώς μπορούν να γίνουν βελτιώσεις στην πολιτική και τέλος πώς αυτές οι πολιτικές θα συνεισφέρουν θετικά στην ε, ανθρώπινη ανάπτυξη και εξέλιξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων έχουμε εστιάσει στη δημιουργία εθνικών πολιτικών για την δημιουργία πρόσβαση στην, στον ε, πολιτισμό. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ισορροπημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες πολιτισμού, βελτίωση της κινητικότητας των καλλιτεχνών, διότι χωρίς αυτούς ποτέ δεν θα μπορέσουμε να επιτεύξουμε τους στόχους μας και πώς μπορούμε να εντάξουμε τον πολιτισμό στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ο πολιτισμός γίνεται όλο ένα και πιο σημαντικό στοιχείο της ε, πολιτικής. Αυτό φαίνεται και ε, σε αυτά που κάνουμε στην ε, UNESCO. Και επίσης να μην ξεχνάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν υπάρχει πολιτισμική έκφραση χωρίς ελευθερία, χωρίς σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης. Και στη δική μας περίπτωση στην καλλιτεχνική ελευθερία και τα δικαιώματα του καλλιτέχνη που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της σύμβασης. Προσπαθήσαμε λοιπόν όλους αυτούς τους στόχους να τους συγκεντρώσουμε, να τους πλαισιώσουμε και αναπτύξαμε ένα σύστημα δικτών. Είναι ένα πολύπλοκο, δύσκολο και ε, καθόλου οικονομικό σύστημα. Ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτό το σύστημα δικτών, έτσι ώστε να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα, το πόσο αποτελεσματικές είναι οι πολιτικές μας. Αυτό που κάναμε είναι να συγκεντρώσουμε αυτούς τους τέσσερις στόχους, να τους χωρίσουμε σε δέκα επιμέρους τομείς και να ε, έχουμε εμπειρογνώμονες για τον κάθε τομέα. Την, ε, προσεχώς θα έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε ε, τα στατιστικά στοιχεία που θα προκύψουν από αυτούς τους δείκτες και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να γίνει αυτό το σύστημα ο τρόπος μέτρησης των ε, αποτελεσμάτων της πολιτισμικής πολιτικής. Πηγαίνουμε λοιπόν προς αυτήν την κατεύθυνση. Είμαστε δηλαδή, έχουμε δράσει με καινοτόμο τρόπο Πιστεύω, ανταποκριθήκαμε στην πρόκληση που μας ετέθηκε, γι' αυτό χρειαζόμαστε όλη τη στήριξη που μπορούμε να έχουμε. Το 2015 άρχισε η εξέταση για την, έκθεση που, για την νομοθεσία που θα εφαρμοστεί από το 2017 και μετά. Τώρα, τι βρήκαμε στην έκθεση, στις αρχικές εκτιμήσεις μας. Κάποιους στόχους, ε, στόχο οι πολιτικές πρέπει να βασίζονται σε διαφάνεια. Και τι αποτελέσματα έχουμε δει μέχρι τώρα. Ότι, οι, ότι έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία 10 χρόνια πολιτικές ε, για τον πολιτισμό, ταυτόχρονα όμως λείπει ένα σύστημα παρκούς αξιολόγησης των εξελίξεων. Επίσης, η κοινωνία των πολιτών παίζει πάρα πολύ σημαντικό ε, ρόλο ως ε, θεματοφύλακας αυτών των εξελίξεων, όμως αυτή τη στιγμή δεν στηρίζεται αρκετά. Χρειάζεται λοιπόν να δοθούν περισσότερα ε, κίνητρα και να δημιουργηθούν περισσότερες ε, συνέργειες. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρούμε απαντήσει σε αυτές τι ερωτήσεις. Τώρα, δεύτερο στόχο, ομαλή ε, ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Εδώ έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να καταλήξουμε σε ένα ομαλό σύστημα ανταλλαγής ε, πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών η παγκόσμια αγορά είναι τεράστια και εξελίσσεται ταχύτατα. Νομίζω πως ε, εξελίσσεται με, ταχύ, με τους ε, ταχύτερους ρυθμούς από όλες τις υπόλοιπες αγορές. Μόνο η Κίνα και η Ινδία αποτελούν το 20%. Μάλλον, αν εξαιρέσουμε την Κίνα και την Ινδία, το 20% των ε, πολιτισμικών αγαθών δημιουργούνται και ε, καταναλώνονται από αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε με ε, προσοχή για να δούμε και τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν και πώς θα λυθούν αυτά. Επίσης, οι νέες εμπορικές συμφωνίες και το πώς το πλαίσιο αυτό επηρεάζει τον πολιτισμό. Τρίτος στόχος. Ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης και των αναπτυξιακών στόχων και των στόχων μάλλον της χειριτής τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εδώ πιστεύω πως ε, απέχουμε πολύ από το να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Είχαμε αρκετούς οικονομικούς περιορισμούς Μειώνονται, μειώνεται η χρηματοδότηση. Το 2008 είχαμε 1%, τώρα έχουμε 0,8%. Έχουμε χάσει δηλαδή αρκετά. Και όπως έχετε παρατηρήσει και εσείς με την ιδιότητα της Πρόεδρου αυτής της Επιτροπής, κάθε, ε, όταν μάλλον πρέπει να γίνουν περικοπές κάπου, πρώτα αρχίζουν από τον πολιτισμό. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα η πρόθεση δηλαδή, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των ελευθεριών που υφίστανται επιθέσεις απανταχού του κόσμου. Το 2004, 237 επιθέσεις κατά των ε, δικαιωμάτων της ε, έκφρασης σε πάρα πολλές δεκάδες χώρες. Πολύ ε, σημαντικά πράγματα, δηλαδή μιλούμε για για λογοκρισία σε βάρος ε, δημιουργών κλπ. Και περιορισμό βέβαια της καλλιτεχνικής έκφρασης, πάρα πολύ ε, σημαντικό και με σημαντικές οικονομικές απώλειες, άρα δεν είναι καθόλου καλή η κατάσταση στον γύρο αυτό και ε, μάλιστα χειροτερεύει. Πρέπει επίσης να σημειώσω την έλλειψη ισότητας ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες εκπροσωπούνται πολύ περιορισμένα σε έναν αριθμό επαγγελμάτων που έχουν σχέση με την καλλιτεχνική έκφραση και ε, για να ολοκληρώσω σιγά σιγά την παρουσίασή μου, έχω και ορισμένες συστάσεις, βασικές συστάσεις δηλαδή της εκθέσεώς μας. Και πρώτα, σημειώσαμε εδώ και μια δεκαετία περίπου ότι ανοίγουν νέοι τομείς εργασίας που θα πρέπει να περιληφθούν στην σύμβαση ορισμένες από αυτές, διότι αλλιώ η πολιτιστική πολυφωνία δεν μπορεί να προστατευτεί. Θα ήθελα να τονίσω ε, και τα δημόσια μέσα και τις ψηφιακές τεχνολογίες είναι δύο τομείς όπου επιθυμούμε να συνεχιστεί ο προβληματισμός και η δραστηριότητα της ε, συμβάσεως διότι εάν δεν διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή της συμβάσεως θα αποτύχουμε. Πρέπει να περιλάβουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ε, διακυβερνητική συνεργασία γιατί είναι πολύ σημαντική τομή αυτή για να μπορέσουν με τη βοήθειά τους να υλοποιηθούν οι στόχοι της συμβάσεως. Το άλλο είναι η ροή των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, προτιμησιακά ε, μέτρα για την στήριξη των καλλιτεχνών και προώθηση μιας πιο ισορροπημένης ροής πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, επίσης η αηφόρος ανάπτυξη, ο πολιτισμός πρέπει να μπει στην καρδιά αυτών των στρατηγικών αηφόρων αναπτύξεως. Είναι και εργαλείο και για την ανάπτυξη ειρηνικών κοινωνιών συμφιλίωση. Είναι πολύ σημαντικά τα πράγματα αυτά στο σημερινό κόσμο. Και τέλος, η προώθηση του ρόλου των γυναικών. Διότι οι γυναίκες είναι και αυτές που παράγουν περισσότερο πολιτιστικό περιεχόμενο. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την παρακολούθηση αυτή, το monitoring δηλαδή, έχουμε και έναν αριθμό περιοδικών εκθέσεων, ζητώ συγγνώμη κάπως μακριγόρο τώρα, είναι οι βασικές πηγές πληροφοριών μας και είναι εκθέσεις που ε, εκδίδουν οι χώρες μέλη, τις δημοσιεύουμε και στην ιστοσελίδα μας. Βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παράγει, δηλαδή συντάσσει τέτοιες εκθέσεις. Στον πρώτο αυτόν κύκλο του monitoring διαπιστώσαμε ότι έχουν εμφανιστεί πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα από αυτά. Μια και νομίζω ότι είναι σημαντικά για σας που ε, διαμορφώνετε την ευρωπαϊκή πολιτική. Και πρώτα η ευρωπαϊκή ατζέντα πολιτισμού. Συμβαδίζει απολύτω με το περιεχόμενο τη συμβάσεω, προωθεί ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδει ελευθερίε, πολιτιστική πολυφωνία, τον διαπολιτιστικό διάλογο που είναι καταλήτη τη δημιουργία. και βεβαίω παίζει σημαντικό ρόλο και στι διεθνεί σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Επίση τα διάφορα ε, πρωτόκολλα για πολιτιστική συνεργασία τα οποία έχει συνυπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, 7 ε, ε, ε, συμφωνίες με χώρε όπω η Γεωργία, ο Καναδά και άλλε. Πολύ σημαντικέ αυτέ και διασφαλίζουν και μια συνέχιση τη προσπάθεια αυτή, γιατί είναι σωστό τρόπο για να αντιμετωπίσουν τα πράγματα αυτά, ενισχύουν και τη σύμβαση, ενισχύουν και το έργο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το άλλο θέμα τώρα είναι το ζήτημα της ατζέντα της ψηφιακής τεχνολογίας που ε, ιδρύθηκε το 2007 και ε, που η ε, ψηφιοποίηση αποφέρει πάρα πολύ σημαντικά τεχνολογικά και εμπορικά ωφέλη. Έχουμε επίσης τα εργαλεία γεωγραφικής συνεργασίας για να μπει ο πολιτισμός στο πλαίσιο της ε, βιώσιμης αναπτύξεως. Έχει μπει τώρα η Ευρώπη στο δεύτερο κύκλο, έχει συνταχθεί το πρόγραμμα της Ευρώπης, το Euro Program. Δηλαδή, νομίζω λοιπόν με λίγα λόγια ότι ως ευρωβουλευτές, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παίζεται ένα σημαντικό ρόλο για την πρόθεση όλων αυτών των διαδικασιών. Έχουμε την εφαρμογή του άρθρου 16 της συμβάσεως που εξασφαλίζει την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών και το 21 της ε, Συμβάσεως για Διεθνείς Συνεργασίες που ε, ζητεί από τις χώρες μέλη να αναλαμβάνουν τις ευθύνες για την προώθηση των στόχων της Συμβάσεως και σε άλλα διεθνή βήματα, φόρουμ δηλαδή. Ε, παίζεται σημαντικό ρόλο, παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σημαντικό ρόλο και σας ευχαριστώ για αυτό. Υπάρχουν αυτά αποτελέσματα λοιπόν, νέες πολιτικές, νέα νομοθεσία σε πολλές χώρες μέλη και ούτω Βεβαίως οι ευρωβουλευτές μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα για να στηρίξουν αφήνω εκτός το θέμα του προπολογισμού που βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Εσείς είστε οι διαχειριστές του προπολογισμού αλλά με την νομοθεσία, με την τροποποίηση των υφισταμένων νόμων μπορείτε να ενισχύσετε πολύ το έργο της συμβάσεως. Ακόμα και οι συζητήσεις περί πολιτικής, ε, στα θέματα αυτά δηλαδή, θέτουν τα ζητήματα του πολιτισμού, ε, βεβαίως μέσα από το κοινοβουλευτικό σύστημα και σε αυτό συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο το δυνατόν περισσότερο. Και τέλος και η ε, διασπορά, η διάδοση και μετάδοση του κειμένου της συμφωνίας και σε άλλες συμβάσεις δηλαδή και σε, άλλους, και σε άλλες γλώσσες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ρόλο καταλήτη για να εξασφαλιστεί μια μεγαλύτερη ορατότητα τη συμβάσεως. Και εμεί παίζουμε το ρόλο μας. Ενισχύουμε τι κυβερνήσει, στη συλλογή δεδομένων. Δεν θα το συζητήσω περισσότερο αυτό. Ε, διαμορφώνουμε και ενότητες εκπαιδεύσεως που μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες μέλη για να βελτιώσουν το policy making προσφέρουμε και χρηματοδοτική υποστήριξη μέσω των κονδυλίων που μπορούμε να αντλήσουμε από διάφορες πηγές. Αυτό, η έκθεση αυτή συντάχθηκε ήδη και εκδόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Ήδη εμπνέει τις κυβερνήσεις τη διαμόρφωση των πολιτιστικών πολιτικών τους και από την Ινδονησία μέχρι την Νότια Αφρική. Έχουμε 144 χώρες μέλη και πάνω από 100 μας προσφέρουν ενίσχυση και δεδομένα τα οποία και εμείς μεταδίδουμε στο κοινό. Σχεδιάζουμε τώρα μια δεύτερη έκδοση της εκθέσεως για του χρόνου. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και μάλιστα να την παρουσιάσουμε και μαζί σας. Θα ήθελα τελειώνοντας να ευχαριστήσω και εσάς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της για την υποστήριξη που έχουμε λάβει. Και είμαστε εδώ και η μου και εγώ για να απαντήσουμε σε ενδεχόμενες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση σας και πραγματικά πηγή ε, εμπνεύσεως για μας. Πολύ σημαντική η πολιτιστική πολιτική της UNESCO και βεβαίως η συνεργασία που έχουμε μαζί σας και ούτως ή άλλως αλλά και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Θα συνεχίσετε τελικά. Λοιπόν, θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν παρεμβάσεις από πλευρά συναδέλφων για την παρουσίαση. Η κυρία Τρούπελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Σίλβια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Αναφερθήκατε στην ε, ε ειδική μεταχείριση, προτιμησιακή μεταχείριση και αναφερθήκατε και στις ε, διεθνείς συνθήκες. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω, διότι τώρα ε, ξέρουμε ότι στις διαπραγματεύσεις για την TTIP οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν κύρωσαν τη σύμβαση ε, αλλά ο Καναδάς την κύρωσε. Επομένως θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον έχετε κάποια αξιολόγηση για την συμφωνία με τον Καναδά, τη ΣΥΤΑ, για τον πολιτισμό και το πολιτιστικό περιεχόμενο και αν στο παρελθόν είχατε καμία σχέση με αυτούς οι οποίοι διαπραγματεύτηκαν αυτές τις ε, συνθήκες. Σας ζητούν ε, να δώσετε συμβουλές, να γνωμοδοτήσετε. Υπάρχει καμία σχέση με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κυρώσει τη σύμβαση. Υπάρχει σχέση μεταξύ των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ε, ημών. Θα συλλέξουμε πρώτα τις ερωτήσεις. Ε, θέλει κανείς άλλο το λόγο. Κανείς. Πριν ε, δούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο που θα θέλει το λόγο, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Εσεί γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν υπόδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκίνησε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση με μια πολιτιστική διπλωματία, αν θέλετε, παρόλο που έχει και πολλά άλλε διακλαδώσει. Ε, ο πολιτισμό, λοιπόν θα πρέπει να ε, αφορά τι ε, διεθνεί σχέσει τη ευρωπαϊκή Ένωση. και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική και η συνεργασία με την UNESCO για αυτή την πολλά υποσχόμενη νέα στρατηγική που είναι και μια στρατηγική ειρήνη. και επειδή μα ασχολούν και τα θέματα της Ευρωμεσογείου, θα ήθελα να ξέρω αν σκοπεύετε να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή την ε, νέα πιο ολιστική προσέγγιση, γιατί και η υπατή η κυρία Μογκερίνη, αλλά και ο αρμόδιος επίτροπος ε, για θέματα παιδείας και πολιτισμού και τα θέματα πολιτικής γειτονίας μας απασχολούν εδώ. Δεύτερον, ελευθερία και καλλιτέχνες, επιθέσεις προς τους καλλιτέχνες και ελευθερία της εκφρασής τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα εμείς το συζητήσαμε και με τις διάφορες πολιτικές ομάδες και θα γίνει και μια συζήτηση που αφορά το θέμα της ελευθερίας της έκφρασης και των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης, αλλά πιστεύω ότι αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο και θα ήθελα να ξέρω και αν υπάρχουν κάποια στοιχεία στην έκθεση. Θα μπορούσαμε να το ε, να στο θέμα αυτό σε Επιτροπή Πολιτισμού και να υπενθυμίσω ότι ε, στο θέμα των προξενικών θεωρήσεων ε, είναι περιορισμένες οι δυνατότητες που έχουμε. Ναι, μεν ε, για την Ευρώπη, για τους καλλιτέχνες έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες για περιοδίες, θειάσους που εμφανίζονται σε κάποιες περιοχές κλπ. Και υπάρχει κανονισμό που προβλέπει για ερευνητές, ε, για διδάσκοντες, ε, φοιτητές ε, και καλλιτέχνες κάποιες δυνατότητες να κυκλοφορούν καλύτερα υπήκοοι τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πια μεγαλύτερε ευκολίες πρόσβασης. Εξακολουθεί να μας απασχολεί το ζήτημα. Και επίση είναι και πάρα πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον που δείχνεται για του δείκτε για τον πολιτισμό. Σω δεν το γνωρίζετε, αλλά έχουμε ζητήσει από την αρμόδια γενική διεύθυνση να εμβαθύνουμε στο θέμα των ε, δικτών πολιτισμού, γιατί εμείς έχουμε αυτό το θέμα. Γίνονται περικοπές στον πολιτισμό, ε, είναι μόνο για περιόδους όπου είναι παχές οι αγελάδες ε, και όταν υπάρχει οικονομική κρίση περικόπεται ο προπολογισμό. Επομένως υπάρχουν ωφέλη που έχει ο πολιτισμός, δεν είναι μόνο οικονομικής φύσεως, αλλά βοηθούν στη συνοχή, υπάρχει δημιουργικότητα του κλάδου αυτού. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο μας αποσχολεί και θα θέλαμε να ξέρουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε επ' αυτού, διότι και εμείς ε, στο θέμα αυτό, ε, στα πλαίσια της Δημιουργικής Ευρώπης, έχουμε ζητήσει μια μελέτη σκοπιμότητας, η οποία υλοποιήθηκε και συνεχίζουμε από αυτό και θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνεργασία. Δεν λέω άλλα για να μην μακρηγορήσω και θα σας δώσουμε λοιπόν αυτά τα λίγα λεπτά για να απαντήσετε αν δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω καταρχάς στην ερώτηση για το εμπόριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και στρατηγικά τα θέματα αυτά. Αν δεν υπάρχει μια κατάλληλη πολιτική από αυτόν, τα υπόλοιπα δεν έχουν και καμία συνέπεια. Όπως είπατε, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν συμμετέχουν σε αυτή τη σύσμαση και μάλιστα ήταν και αντίθετοι στην ε, δημιουργία αυτή της σύμβαση ε, και καταψήφισαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούν τη σύμβαση. Αντιθέτω, παρακολουθούν τη σύμβαση. Διότι είναι μια χώρα με τεράστια κολοσιαία συμφέροντα. Επομένως, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, συμμετέχουν άμεσα υπό την έννοια ότι παρακολουθούν την εφαρμογή της σύμβασης, αλλά δεν την έχουν κυρώσει. Αυτή τη στιγμή η σύμβαση δεν έχει ξεκινήσει συζητήσεις για μεγάλες ε, εμπορικέ συμφωνίε. Δεν έχουν τεθεί μάλλον στη συζήτηση τα θέματα τη σύμβαση. Αλλά τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να το κάνουν αυτό και τα επόμενα χρόνια θα αναπτύξουν ένα πρόγραμμα για εμπορικέ διαπραγματεύσει. Προβλέπεται αυτό για το 2017, διότι σαφέστατα τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή που υπάρχει πλέον μια κρίσιμη μάζα μελών στη σύμβαση, αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για ένα ε, πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο και θα μπορούσαν να συζητηθούν οι αρχές της στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Χρειαζόμαστε βέβαια και τη στήριξη των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά μόνοι μας. Ορισμένες φορές ε, η UNESCO θεωρείται κάτι σαν Σούπερμαν που μπορεί να παρέμβει παντού. Αλλά εμείς είμαστε ένα τίποτα χωρίς τα κράτη-μέλη. Επομένως, ε, χρειαζόμαστε την υποστήριξη των κρατών μελών και την υποστήριξη προς την UNESCO για να μπορέσουμε να μεταλαμποδέσουμε αυτές τις αρχές. Οι αρχές αυτές αντανακλούν ιδέες τις οποίες υποστηρίζουν οι πάντες. Ελευθερία της έκφρασης, για παράδειγμα. Όλοι την υποστηρίζουν την ελευθερία της έκφρασης. Το πρόβλημα είναι πώς μπορούν να εκφραστούν αυτά ρητός ε, στις εμπορικές συμφωνίες. Αρχίζουμε λοιπόν να εισερχόμαστε σιγά σιγά σε αυτούς τους τομείς. Δεν θα πω ότι είναι εύκολο γιατί παίζονται πολύ μεγάλα συμφέροντα, αλλά γνωρίζω ότι η σύμβαση τώρα που είναι αρκετά ισχυρή και αν τύχει και τις κατάλληλε υποστήριξης μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για να μπορέσει να καθοδηγήσει και κάποιες από τις διαπραγματεύσεις ε, προς τον κοινό μας στόχο. για την ερώτηση τη δική σας, κυρία Πρόεδρε. Ναι, συμμετέχουμε σε πολλές από τις δραστηριότητες, κάποιες αφορούν ε, τη σύμβαση αυτή, κάποιες άλλα πράγματα. Θα είδατε ότι πριν από κάποιες μέρες η UNESCO διοργάνωσε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στις Βρυξέλλες, 9 και 10 Ιουνίου, για την επίθεση στον πολιτισμό και ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα, μια πολύ σημαντική ε, διάσκεψη στην οποία συζητήσαμε ε, αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον πολιτισμό σε περιοχές όπου υπάρχει κρίση, σύραξη, ε, ακόμα και μια περίοδος ένδυας και στέρησης πόρων είναι κάτι το οποίο πλήττει τον πολιτισμό. Η κυρία Μογκερίνη απέστειλε ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα παρεπιπτόντω, παρουσιάζοντα τη νέα πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι σχεδόν θαύμα που αυτή τη στιγμή έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον πολιτισμό. Ε, δημοσιεύτηκε στις 8 Ιουνίου η σχετική ανακοίνωση. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα προς την ε, σωστή κατεύθυνση και θα ήθελα ε, να το αναφέρω ως κάτι το οποίο θα επαναπροσανατολίσει τις ε, θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί και τα Ηνωμένα Έθνη ορισμένες φορές δεν στοχεύουν τόσο καλά και δεν υποστηρίζουν τόσο καλά τις πολιτικές περιπολιτισμού όσο θα έπρεπε. Για μας είναι ένα άλμα προς τα μπρος, ε, ένα γιγάντιο άλμα για τις ε, πολιτικές για τον πολιτισμό. Και φυσικά με βάση αυτό ε, μπορούμε να αναπτύξουμε πολλές άλλες πολιτικές. Προστασία του πολιτισμού, διαπραγματεύσεις σε εμπορικό πλαίσιο, πολιτική προξενικών θεωρήσεων. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι υπάρχει και μια σχετική πρωτοβουλία για διευκόλυνση ε, στις ε, προξενικές θεωρήσεις και πολλά άλλα τα οποία αναφέρατε, δείκτες για τον πολιτισμό κλπ. Αυτά είναι τα όσα θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια. Ε, προσβλέπουμε στην ουσιαστική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το πολύ σημαντικό τομέα πολιτικής. Και πάλι να σας ευχαριστήσω, να υπενθυμίσω ότι θα σας χρειαστούμε διότι θα είμαι και εισηγήτρια για την νέα ανακοίνωση για την πολιτιστική πολυμορφία. Επομένως, εναπόκειται σε μένα να συνεργαστώ μαζί σας και να λάβουμε υπόψη και την πολύ πολύτιμη συνεισφορά σας και Υπάρχει και πιθανό άλλο πεδίο γόνιμη συνεργασίας γιατί καταφέραμε το 2018 να είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ε, είναι λοιπόν ένα ακόμα τομέα στον οποίο θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ λοιπόν και για αυτό το πολύ σημαντικό έγγραφο το οποίο μα αφήσατε, για αυτή την έκθεση και για αυτό το άλλο έγγραφο το οποίο θα διανύμω, ε, θα το συζητήσουμε με τη Γραμματεία, επένδυση στην, ε, στον πολιτισμό για βιώσιμη ανάπτυξη που είναι το αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής έρευνας και θα έχουμε και την έκθεση της Επιτροπής μας με την Επιτροπή Βιομηχανίας για την Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία. Έχετε δίκιο για το θέμα αυτό. Μας απασχολεί ιδιαίτερα η επίθεση στην πολιτιστική κληρονομιά. Θεωρούμε ότι το θέμα των καλλιτεχνών και της ελευθερίας της έκφρασής τους των δημιουργών ε, τους οποίους, στους οποίους επιτίθεται είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να εμβαθύνουμε και θα πρέπει να έχουμε και εμείς την άποψή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Με αυτό ολοκληρώνεται η πρωινή συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε στις 3 η ώρα. Θα έχουμε πρώτα τον Επίτροπο Νευράτσιτς για το θέμα Τη νέα αυτή αφήγηση για την Ευρώπη. Θα έχει μια ανταλλαγή απόψεων από αυτό και ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή, τον κύριο Τάκουλα και ε, τους κοιόδης για τι πολιτικέ για τον αθλητισμό και την παρουσίαση τη μελέτη ε, για τη διπλή ε, ε, καριέρα στον αθλητισμό. Θελήσαμε να συνδυάσουμε τα δύο αυτά τα θέματα. Ελπίζω να υπάρχει παρουσία όλων των συναδέλφων και σα παρακαλώ να είστε παρόντες. Θα επανέλθουμε δρυμύτερη στις 3.